Μακλάρκεν και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εστιάσουμε σε τρία από τα τέσσερα βασικά στοιχεία του προγράμματος πλαισίου που είναι τα κέντρα αριστείας και οι προκλήσεις της ε, κοινωνίας. Εγώ, σαν μέλο τη Επιτροπή Περιβάλλοντο, γνωρίζω πολύ καλά ποιε είναι οι προκλήσει οι οποίε αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και ιδίω τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή και τη δημόσια υγεία. Και χαίρομαι που ένα μεγάλο τμήμα του προπολογισμού μα θα αφορά έρευνα στα θέματα αυτά. Θα ήθελα να εξασφαλίσω ότι ο προϋπολογισμός της Κομισιόν δεν θα υποστεί περικοπές στις διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία αυτού του προϋπολογισμού και να θέσουμε το Κοινοβούλιο σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση και να εξασφαλίσουμε ότι θα διατηρηθεί το ποσό που προτείνει η Κομισιόν. Είναι θετικό να υπάρχει και εμνία για την έρευνα για τα πολιτιστικά θέματα και την πολιτιστική πληρονομία που έχει δοθεί <clears throat> στην πολιτιστική κληρονομιά προτεραιότητα από την Κομισιόν που είναι κάτι το σημαντικό για το νέο πρόγραμμα. Η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη για να μην εξαλειφθεί το θέμα αυτό από μελλοντικέ προτάσεις στο πρόγραμμα πλαίσιο. Όπως ξέρετε υπάρχει μια αναφορά η οποία ζητά να υπάρξει προστασία της πολιτικής κληρονομιάς των ορίζον 2020, γιατί έχει μια βασική αξία πνευματική αλλά και οικονομική, όχι μονάχα για τον τουρισμό, αλλά επίσης και για να ενθαρρύνει την δημιουργικότητα και να δώσει έμπνευση για περαιτέρω καινοτομία. Όπως είπα και σε μια προηγούμενη ευκαιρία, θα πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στη γνωμοδότηση αυτή ο ρόλος της κουλτούρας και της πολιτιστικής πληρονομιάς, όπως και στα προηγούμενα προβλήματα. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί η σημασία <clears throat> της σωστής επιλογής των επιστημονικών προγραμμάτων και να δοθεί έμφαση στο ρόλο των γυναικών στην επιστήμη, ώστε περισσότερες γυναίκε να συμμετέχουν στην επιστημονική δραστηριότητα και να έχουν είδε ευκαιρίες και να έχουν ίση υποστήριξη στον τομέα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση, εάν μας ενδιαφέρει, να μεγιστοποιήσουμε την καινοτομία. Επίσης για τα επιστημονικά θέματα πρέπει να υπάρξει κίνηση από την παλιά προσέγγιση να έχουμε πόλους αριστείας σε συγκεκριμένα μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βελτιώσουμε αντίθετα την κατάσταση σε όλα τα ερευνητικά κέντρα. <clears throat> Από τη δική μου πλευρά, ω σοσιαλίστρια, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ίση χρηματοδότηση σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το να συνδυάσουμε τι προτάσει του Horizon 2020 μαζί με τα τμήματα που αφορούν την καινοτομία στο Ταμείο συνοχή με τη δημιουργία ικανότητα η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αριστεία. Με τον τρόπο αυτό τα κράτη-μέλη, τα τμήματα των κρατών μελών που υπολείπονται στα επιστημονικά του προγράμματα μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητά του και να μπορέσουν έτσι να υποφελθούν πλήρω του προγράμματο Horizon 2020. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να επωφεληθεί γενικότερα με το να έχει περισσότερες επιστημονικές προοπτικές και περισσότερη δυνατότητα καινοτομία και πάλι καλωσορίζω την πρόταση της Emma και ε, προσβλέπω σε καλή συνεργασία με την εισηγήτρια και τους άλλους σκιώδες εισηγητές για το Ροΐζον 2020. Ο λόγος τώρα στον κύριο Μπόρις. E, e, Ευχαριστώ και εγώ ε, συμφωνώ με την κυρία Μακλάρκιν. Στις περισσότερες από τις προτάσεις της. Και εγώ έχω συντάξει τρεις γνωμοδοτήσεις στην Επιτροπή Γιούρε. Ε, μερικά σημεία είναι ταυτόσιμα, Ωστόσο, στο πλαίσιο της εκπαίδευση θα ήθελα να προσθέσω ότι κάτι δεν ήταν σημαντικό είναι ότι στον, ε, στο σχέδιο του Ορίζον 2020 υπάρχει μια συνέργεια με το πρόγραμμα Erasmus for All για όλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, σημείο γιατί έχουμε και την κινητικότητα των ε, των φοιτητών διδακτορικού τίτλου και των κατόχων διδακτορικού τίτλου, κάτι το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε όλα τα επίπεδα, ε, όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει και μια συνέργεια μεταξύ του προγράμματος Horizon 2020 και Εράσμους για όλους. Δεύτερο σημείο ε, για την αριστεία στην επιστήμη. Θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της επένδυσης στην επιστημονική έρευνα. Πρόσφατα εγκρίναμε πολλές ε, γνωμοδοτήσεις ε, και εκθέσεις για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δυστυχώς, οι ενέργειες που αναλαμβάνονται για την στήριξη προς τη διδακτική και ε, ερευνητική βάση, εντάξει, έχουμε κάνει κάποια βήματα, αλλά πρέπει να τα βελτιώσουμε ακόμα περαιτέρω ούτω ώστε τα πανεπιστήμια να είναι σε θέση να αξιοποιούν τα κονδύλια αυτά για την βελτίωση της διδακτικής τους βάσης. Τρίτο σημείο, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο εξή. Στον αντίκτυπο του ορίζον 2020 στις τρίτες χώρες και στην πολιτική γειτονία. Όπως και το Erasmus Mundus, το πρόγραμμα Marie Curie και αυτό θα πρέπει να ε, τα λαμβάνει όλα αυτά υπόψη. Να υπάρχει λοιπόν αναφορά και στην πολιτική, στην πολιτική γειτονίας, αλλά και στην αναγνώριση των ε, ε δεκτορικών ε, τίτλων. Χαίρομαι που στο μέλλον το πρόγραμμα Marie και ως Πολωνός χαίρομαι που το στο όνομα Marie θα προσθέσουμε και το ε, καταρχικό της όνομα Ποτροσκόφσκα. Είναι συμβολική η αξία, αλλά για μένα είναι σημαντικό. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι η στήριξη στο τρίγωνο της γνώσης. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας, ε, που θα αντλήσει πολλά από αυτά τα κονδύλια, θα, θα ε, μπορεί έτσι να έχει και σε πρακτικό επίπεδο συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Καταδεικνύοντας ότι η έρευνα ε, στα πανεπιστήμια στη συνέχεια θα μεταφερθεί και στην ε, οικονομία. Προηγουμένως δεν υπήρχε αυτή η άμεση σύνδεση. Και το τελευταίο που θα θέλω να αναφέρω είναι κάτι που χρηματοδοτείται για πρώτη φορά εδώ πέρα. Ε, ε τα, προγράμματα, τα ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τι ανθρωπιστικέ επιστήμες. Αν δείτε τι κοινωνικέ προκλήσεις που είναι ο τρίτο πυλώνας, Πολλέ από αυτές τι προκλήσεις αφορούν την υγεία, τα ενεργειακά συστήματα, τις μεταφορέ, μεταφορές, ε, ε, την ασφάλεια τροφίμων και γενικώ την ασφάλεια θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν και άλλοι τομεί, όπω και οι τομεί των ανθρωπιστικών επιστημών, και εκεί πέρα μπορεί να υπάρξει καινοτομία, και ότι εξάλλου θα πρέπει να λαμβάνεται αυτό υπόψη, αυτή η πτυχή, σε όλε ε, τι ε, δραστηριότητε. Γιατί υπάρχουν πολλά ωφέλη στην καινοτομία στι ανθρωπιστικέ επιστήμε. Όχι μόνο, μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στι ανθρωπιστικέ επιστήμε θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Μαζί με την Emma Μακλάρκιν σίγουρα θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και θα συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Παλιαδέλη. σε όλους. Ε, νομίζω ότι συμπίπτουμε απόλυτα ε, με τους προλαλήσαντες σε ό,τι αφορά και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι οι ανθρωπιστικές σπουδέ ε, ως κομμάτι ε, του μέλλοντος της Ευρώ, Ευρώπης πέφτουν ε, από όλους τους συζητητές ως αναγκαία ε, ο αναγκαίος όρος να περιληφθούν σε αυτό το φιλόδοξο στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας και τεχνολογίας. Να ομολογήσω ότι η καινοτομία δύσκολα ερμηνεύεται, μπορεί να έχει εφαρμογή, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση, με τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Και αυτός ο όρος συχνά αποθαρρύνει τους όσους υπηρετούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους κοινότητες γνώσης καινοτομίας και τεχνολογίας ε, ε, με αποτέλεσμα να μην, παίρνουν, να μην μετέχουν σε διεκδίκηση προγραμμάτων παρά μόνο μέσα από τη διεπιστημονικότητα. Από ίδια πείρα διαπιστώνω ε, με την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για, ακόμη και για προγράμματα στα οποία υπάρχει μια διεπιστημονική διάσταση να διεκδικήσουν χρήματα από τομείς, από, από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανθρωπιστικές σπουδές μοιάζει να μην είναι κομμάτι της έρευνας και σαφώς δεν μοιάζει να είναι κομμάτι της καινοτομίας τουλάχιστον με την τρέχουσα σημασία του όρου. Αυτό, γι' αυτό κάτι πρέπει να κάνουμε. Έχω ήδη υποβάλει μία ερώτηση στην Επιτροπή με ποιο τρόπο προ, προτίθεται να λύσει τέτοιου ζητήματα τα οποία αφορούν στην πολιτική κληρονομιά. Και με αυτό δεν εννοώ μόνον τη φιλολογία, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, αλλά εννοώ την υποστήριξη δραστηριοτήτων όπως είναι οι πανεπιστημιακές ανασκαφές, οι οποίες είναι ένα τεράστιο κομμάτι ε, από το οποίο προκύπτουν νέα στοιχεία για την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και οι οποίες δυστυχώς, το ξέρω από τη χώρα μου, δεν έχουν καμιά απολύτως χρηματοδότηση επειδή ως πολιτιστική κληρονομιά το πακέτο πάει όλο ε, στο Υπουργείο Πολιτισμού και οι πανεπιστημιακές ανασκαφές ανήκουν, στα, ε, ανήκουν, ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Επομένως πρέπει να δοθούν στις ανθρωπιστικές σπουδέ που κάνουν έρευνα η οποία ε, καλύπτεται απολύτως από αυτή τη διατύπωση στο στρατηγικό θεματολόγιο της καινοτομία για μια Ευρώπη με αποδοτική χρήση των πόρων της. Γιατί εκτιμώ ότι ένας από τους μέγιστους πόρους της Ευρώπης είναι η πολιτιστική της κληρονομιά. Γι' αυτό έχουμε υποχρέωση με κάθε τρόπο να τη στηρίξουμε αυτή την ε, διάσταση παρά, να τρέχουμε καμιά φορά πίσω από τεχνολογικές αναζητήσεις για τις οποίες άλλοι από άλλες ε, υπήρους έχουν βρει ε, καλύτερους τρόπους. Έχουμε κάτι το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν θέλει και πάρα πάρα πάρα πολλά χρήματα. Ε, συμφωνώ απόλυτα με όσους ε, ε, συναδέλφους μίλησαν προηγουμένως αυτό που δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν προβλέπεται στο στρατηγικό πλαίσιο η συνεργασία με, το, με, το, την Ευρωπαϊκή Περιοχή Έρευνας European Research Area δεν ε, αναφέρεται καθόλου στο, στο κείμενο στην ε, αιτιολογική έκθεση της, για την τροποποίηση του πλαισίου. Θα πιστεύω λοιπόν ότι και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προσθεθεί μια τέτοια διατύπωση. Έχω μια ερώτηση, <coughs> συγγνώμη, την οποία ε, δεν ξέρω αν μπορεί να μου την απαντήσει κανείς σήμερα. Δεν καταλαβαίνω την ίδρυση του Ιδρύματος ε, ε Ευρωπαϊκής ε, του ΕΙΤ. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Τι, τι ρόλο παίζει πέρα από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας δοθεί μια απάντηση αν είναι πραγματικά παραγωγικό. Γιατί αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που κάνει είναι η επικοινωνιακή πολιτική, ενδεχομένως και μια αξιολόγηση. Αλλά ειλικρινά ομολογώ ότι δεν ξέρω πολλά πράγματα για αυτό το ίδρυμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινοτομία και Τεχνολογία και επομένω πρέπει να το ξαναδούμε. Μήπω δηλαδή φεύγουν πόροι οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ε, ακόμη περισσότερο χωρί ένα, ε, ένα νέο θεσμό ο οποίο ε, ενδεχομένω τρώει χρήματα. Ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε με τους ε, εισηγητές προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι σίγουρη, αφού έχουμε τέτοια ομοφωνία σε ό,τι αφορά την πολιτική κληρονομιά και τις ανθρωπιστικές σπουδέ, ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε ώστε οι ανθρωπιστικές σπουδέ να καθιερωθούν ως κομμάτι της επιστημονικής έρευνας και όχι απλό και της καινοτομίας ενδεχομένως, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Κώστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημερίζομαι όσα είπαν οι συνάδελφοι, οι συγγήτρια, αλλά και η κυρία Παλιαδέλη. Νομίζω ότι η Επιτροπή Πολιτισμού θα έπρεπε να υπερκεράσει τις ε, διαφορές γνώμης που υπάρχουν και να λάβει μία θέση απέναντι σε όλα τα άλλα προγράμματα. Γιατί είδα αξιολογώντας το ορίζοντα και όλα τα άλλα προγράμματα ότι η διάσταση του πολιτισμού ε, σιγά σιγά χάνεται στην πραγματικότητα και αυτό είναι πολύ άσχημα. Αλλά και η πολιτική συνοχής, η οποία θα έπρεπε και εκείνη να λάβει περισσότερους πόρους. Τώρα, όσο αφορά τον ορίζοντα, η νέα τριμερής κατανομή στου τρεις πυλώνες που υπογράμμισε και η συγγήτρια, η αριστεία, η βιομηχανική ηγεσία, οι προκλήσεις της κοινωνίας, στο, στο πρώτο δεν γίνεται καμία αναφορά ε, ούτε στα υλικά, ούτε στις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα, ε, μόνο περιθωριακές αναφορές. Στο δεύτερο πυλώνα και πάλι πρακτικά δεν υπάρχει καμία αναφορά και στο πλαίσιο της έρευνας, μόνο εκεί αναφέρεται η πολιτιστική κληρονομιά. Σας θυμίζω σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα, το ενισχύει, στην πραγματικότητα είχε προβλεφθεί ένα ολόκληρο πρόγραμμα ε, για, τον ευρωπαϊκό, για την ευρωπαϊκή κληρονομιά με χρηματοδοτήσεις, πόρους, συγκεκριμένα για την αξιοποίηση, διάδοση και στήριξη της ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς. Ε, υπάρχουν και πολλές συγκεκριμένες αναφορές στην πολιτιστική διάσταση και δια, ε, στον διαπολιτιστικό, διεπιστημονικό χαρακτηριστικό χαρακτήρα της έρευνας. Στο κλείσιμο τώρα ε, του προγράμματος και σε σχέση και με την πολιτική, σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας, θα πρέπει να υπάρξει μία ύπαρξη της συνιστώσας πολιτισμού σε όλες τις πολιτικές μας. Ε, έχουμε λοιπόν και μια νομική βάση. Είμαστε εξοπλισμένοι τώρα. Πιστεύω ότι ε, επίσης το θέμα της ψηφιοποίησης ε, η στήριξη στις τεχνολογίες λοιπά... Μερικές φορές επικαλύπτει, τα επικαλύπτει όλα η ψηφιακή ατζέντα, το ψηφιακό θεματολόγιο και νομίζω ότι έτσι υποφέρει λίγο το μέσο της πολιτισμικής κληρονομιάς. Ε, σε όλα μας τα έγγραφα και κείμενα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την πολιτιστική ε, ένταξη ε, στις χωροταξικές πολιτικές μας παντού, παντού, στα έργα, στα δημόσια και σε όλες εκείνες τις δράσεις που ίσως εκ πρώτης όψεως φαίνονται εξωτερικές προς το πρόγραμμα Ορίζοντας. Ε, πραγματικά θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια να ε, σημειώσει αυτήν την ανησυχία που έχει εκφραστεί πολλές φορές στην Επιτροπή μας δεδομένου του ότι εδώ μιλάμε για 80 δισεκατομμύρια ευρώ, πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις ε, δηλαδή αυτή η αύξηση τα 50 στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, θα ήταν παράξενο να μην βρεθεί μια θέση για την πολιτιστική διάσταση της έρευνας, που μπορεί επίσης να δώσει και μια όθηση στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων πολιτιστικών επιχειρήσεων. Στον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ποτέ δεν μιλούμε για αυτές τις δημιουργικές πολιτιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται. Έχουμε λοιπόν όλο αυτό το προϋπολογισμό των 80 δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων, αλλά τι πάει σε κάθε αποδέκτη είναι πολύ διαφοροποιημένο. Σας ευχαριστώ κυρία Κώστα και τώρα η κυρία Φεράιερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μακλάρκεν και να τη συγχαρώ για την ποιότητα τη εργασία του. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και την πολιτιστική πλευρά και την πλευρά του αθλητισμού στο πρόγραμμα πλαίσιο. Κάτι το οποίο με ικανοποιεί λιγότερα είναι το θέμα αυτό της έρευνας για την πολιτιστική κληρονομιά, για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την τεχνολογική ε, καινοτομία, αλλά όλα αυτά να παρουσιάζονται σαν εναλλακτικέ ή αντίπαλε δυνατότητε. Εγώ νομίζω ότι αντίθετα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διάδραση μεταξύ <clears throat> τη τεχνολογία και των ανθρωπιστικών επιστημών, παραδείγματο χάρη τη πολιτιστική κληρονομιά, γιατί βλέπουμε κάθε μέρα ότι τα μέσα ενημέρωση έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία τη επικοινωνία Όλα αυτά οδηγούν σε νέε προκλήσεις, οδηγούν σε νέε προκλήσει και για τον πολιτιστικό τομέα και κατά την άποψή μου υπάρχει πολύ λίγη έρευνα σε σχέση με τη διαδικτύωση και την αλληλοσύνδεση όλων αυτών των τομέων. Δεν πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό της ε, έρευνας σε ανθρωπιστικό και τεχνολογικό χώρο. <clears throat> Νομίζω ότι η σύμπραξη των δύο αυτών πλευρών δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. Η αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνικής εξέλιξης και τεχνολογικής εξέλιξης έχει ένα σημαντικό ρόλο στην ε, ανθρώπινη δραστηριότητα. Και επομένω, εμεί, σαν Επιτροπή Πολιτισμού, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα αυτό, να δούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η νέα τεχνολογία, ιδίως οι τεχνολογίες των επικοινωνιών στα μέσα ενημέρωσης Και ενώ συγχρόνω θέλουμε να διατηρήσουμε τις ε, συνέπειε που έχουν οι τεχνολογίες στον κόσμο της πολιτιστικής κληρονομιάς και της δημιουργίας πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να αντιδράσουμε εγκαίρως σε προβλήματα όπως τα προβλήματα του copyright και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε με το copyright δείχνουν ότι δεν υπήρξε μια αρκετά πρώιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν από τις νέες τεχνολογίες. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ πολύ. Η ΕΜΑ θεωρώ ότι έκανε μια πολύ καλή σύνοψη του προγράμματος ε, πλαίσιο ε, για τις διάφορες στοιχέ του ορίζοντα 2020 και εστιάστηκε σε αυτούς τους τρεις κύριους πυλώνες. Οι πολιτικέ στοιχέ έχουν σχέση και ορισμένα στοιχεία τη βιομηχανική ηγεσία, αλλά κυρίω πρέπει να εστιαστούμε στι κοινωνικέ ε, αλλαγέ. Και εδώ υπάρχει μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τον ορίζοντα 2020 ε, για την ε, πρόοδο σε όλον αυτό το τομέα. Όλοι οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε σημαντικούς τομείς, όπως βεβαίως η πολιτιστική κληρονομιά, οι γυναίκες και η επιστήμη, αλλά και ο αθλητισμός, όπως αναφέρθηκε. Εδώ νομίζω ότι έχουμε μια ευκαιρία να διεξαγάγουμε πραγματική έρευνα ε, προς όφελος ε, του αθλητισμού και ε, της αθλητικής δραστηριότητα, κάτι το οποίο θα συμβάλλει και στην κοινωνία και για την επίλυση ορισμένων ανισορροπιών στην κοινωνία. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κοινωνική ένταξη, αλλά και σε ό,τι αφορά την υγεία γιατί δίνεται μεγάλη έμφαση στην υγεία. Κάθε μέρα συναντιόμαι με εκπροσώπους ε, των λόμπι ε, για την ε, στήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε αυτό το τομέα. Κάποιες φορές νομίζω ότι είναι μια βιομηχανία από μόνη της. Ενώ εμεί πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα για την πρόληψη. Αν κάνουμε περισσότερα για την πρόληψη, τότε δεν χρειάζεται να χρηματοδοτήσουμε τόσο την εξέβρεση θεραπείων. Πολλά πρέπει να γίνουν λοιπόν για τον αθλητισμό, για την φυσική δραστηριότητα και την συμβολή τους στην κοινωνία. Αφενός έχουμε μια ανάπτυξη της συμμετοχής στο, στην αθλητική δραστηριότητα από τους νέους και αγόρια και κορίτσια ευτυχώς. Από την άλλη όμως έχουμε αύξηση της επαχυσαρκίας, κάτι το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα κάποια στιγμή, ασθένειες, ε, απουσία από το χώρο εργασίας κτλ. Και προσπαθούμε να βρούμε θεραπείες, αλλά εγώ θέλω να ε, εστιάσουμε την προσοχή μας πολύ περισσότερο στην έρευνα για τον αθλητισμό, πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή, ε, την, ένα πιο ενεργό αν θέλετε τρόπο ζωής γιατί ο αθλητισμός συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με την ε, υγεία και μια υγιή διατροφή και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε τις κοινωνικές αλλαγές, την κοινωνική, κοινωνική ένταξη κτλ. Αλλά και το ζήτημα της υγείας, κάτι το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Και να δώσουμε έφαση κυρίως στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία της μιας ή της άλλης ασθένειας. Και σε αυτό συμφωνώ απολύτως να δώσουμε δυνατότητες ε, για την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση, υποψηφιότητες, χρηματοδότηση κτλ. Ε, αυτό βεβαίως θα ε, μας οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις, σε μια πιο παραγωγική κοινωνία, γιατί οι άνθρωποι σε αυτήν την περίπτωση, οι πολίτες, θα ζουν για περισσότερα χρόνια, με περισσότερη υγεία και βεβαίω θα είναι και πιο παραγωγική στην εργασία του. Αυτό ελπίζω να μπορέσουμε να το τονίσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Σάντζεσ Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λειτουργεί, λειτουργεί. Εντάξει, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Έμα Μακλάρκιν για την παρουσίασή της και για το γεγονός ότι έθεσε μια σειρά από ερωτήματα τα οποία είναι τμήμα της εργασίας μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ να θέτουμε ερωτήματα. Εγώ θα ήθελα σταθώ στα θέματα της στρατηγικής και της αποτελεσματικότητας της δράσης μας. Νομίζω πρέπει να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες δράσεις και να συνδέσουμε το στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την ε, καινοτομία και τα υφιστάμενα προγράμματα, τουλάχιστον τα προγράμματα για τα οποία θα χρειαστεί να εργαστούμε στο, να εργαστούμε στο διάστημα 2014-2020. Τα προγράμματα λοιπόν που εμπλέκουν την Επιτροπή μας στα θέματα του πολιτισμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη σύνδεση μεταξύ του στατηγικού πλαισίου, της παιδείας, της βιομηχανίας και επίση θα πρέπει, όπω και σε άλλα θέματα, να εμπλέξουμε και την περιφερειακή διάσταση. Είναι οι περιφέρειε τη Ευρώπη οι οποίε έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ικανότητα ανάπτυξη που έχουν και για την προστασία του περιβάλλοντο. Επίση θα πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη έμφαση στο να βρούμε μια ε, βάση, ένα σημαντικό ε, ε, υπόβαθρο για την αριστεία και προφανώς η Επιτροπή μας θα πρέπει να ασχοληθεί και με τα θέματα της κατάρτισης για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε καλύτερα την καινοτομία στο βιομηχανικό τομέα, θα πρέπει να προετοιμάσουμε αυτούς οι οποίοι θα ξεκινήσουν αυτή την καινοτομία. Από τη μία πλευρά λοιπόν θα πρέπει να ενσωματώσουμε στο πρόγραμμα πλαίσιο τα θέματα τα πολιτιστικά, τις αναφορές στον ε, πολιτιστικό τομέα και την παιδεία και την κατάρτιση και να τονίσουμε την ανάγκη να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ευρώπη, ώστε οι προτάσεις μας να συνάδουν με τις άλλες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζω και πάλι το περιφερειακό τομέα που έχει πάρα πολλά κονδύλια και ένα σημαντικό εργαλείο. Θα πρέπει όμως να ενσωματώσουμε την προβληματική της έρευνας και της ε, τεχνολογικής καινοτομίας σε όλα τα προγράμματα στα οποία έχουμε εργαστεί στην Επιτροπή μας και να τα συμπεριλάβουμε στην δημιουργική Ευρώπη, τον έρασμο για όλους κτλ. Και όπως είπαν και προηγουμένως οι προλαλήσαντες, αυτό θα πρέπει να γίνει σε όλους τους τομείς και στον επιστημονικό τομέα που όπως είπε η Σαμπίνε Φερχέιν αυτός δεν είναι ένας τομέας αντίπαλος της κουλτούρας αλλά ένας τομέας ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στην ε, καινοτομία. Απλώς υπάρχει τάση να προχωρούμε πρώτα στον τομέα των θετικών επιστημών, αλλά υπάρχει και ο τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, ο οικονομικός και κοινωνικός στίβος. Υπάρχει επίσης η ψηφιακή, το ψηφιακό θεματολόγιο, η ανάπτυξη στον τομέα αυτό που αποκτά και μεγαλύτερη σημασία και ο χώρος των δημιουργικών ε, δραστηριοτήτων, των πολιτιστικών αυτών δραστηριοτήτων, αλλά και ο τουριστικός χώρος Εάν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια προσθέμενη αξία σε επίπεδο ευρωπαϊκής Ανταγωνιστικότητα, θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλους αυτούς τους φόρους χωρίς να ξεχάσουμε και την ε, επίτευξη μεγαλύτερη πρόσβαση στην έρευνα και την ανάπτυξη ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολλές φορές όλα αυτά τα οποία προτείνουμε λόγω τη πολυπλοκότητας των προγραμμάτων μα δεν είναι πάντα προσβάσιμα στι μικρότερε επιχειρήσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλέ φορέ τα κονδύλια δεν δαπανώνται όπως πρέπει ή δεν δαπανώνται καθόλου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε όλου σε αυτά τα προγράμματα που υποστηρίζουν τη βιομηχανία. Ευχαριστώ. Τάκουλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Έμα Μακλάρκιν. Τα μενήματα που λάβαμε από ε, την ε, συνεδρίαση των ε, σκιωδών εισηγητών μας δείχνουν ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο και συμφωνούμε. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ορισμένα σημεία για τον ορίζοντα 2020, ίσως όμως να είναι πιο σκόπιμο και φρόνιμο να δημιουργήσουμε ποιοτική προστιθέμενη αξία. Δυστυχώς αυτό δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Έχω όμως ορισμένες παρατηρήσεις να κάνω. Αυτό το πρόγραμμα επιδιώκει ε, την ε, ανάπτυξη περαιτέρω προστιθέμενης αξίας στον τομέα της έρευνας. Και αυτό βεβαίως συνδέεται με τη στρατηγική για το 2020. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η έρευνα και η εκπαίδευση είναι το τομή και αυτό το ξεχνούμε κάποιες φορές. Ενδεχομένως η Επιτροπή μας και η Επιτροπή Ήτρε να πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά αν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε αυτή την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Να υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εμείς ε, παρουσιάζουμε αυτή την ε, ε, έκθεση προς την Επιτροπή Ήτρε και θα πρέπει πράγματι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. αυτό το σχέδιο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ε, χρηματοδοτικά μέσα. Αποτελεί όμως ταυτόχρονα μόλις το 5% της συνολικής χρηματοδότησης στην ε, Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την έρευνα. Έχει όμως ε, πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, μπορεί να προωθήσει πολλά μικρότερα ε, προγράμματα και να διαμορφώσουν μια κρίσιμη μάζα, αν θέλετε, ως, από αυτή την άποψη. Η Επιτροπή πρότεινε χρηματοδότηση 80 δις για τον ορίζοντα 2020. Εγώ όμως ανησυχώ γιατί από το Συμβούλιο μας είπαν ότι ο προπολογισμό θα είναι μόλι 60 δι. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Γιατί έτσι ουσιαστικά θα βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση που βρισκόμαστε και τώρα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Ίσως λοιπόν η προστιθέμενη αξία που αναμένουμε ε, να αποκομίσουμε από τον ορίζοντα 2020 να μην ε, υλοποιηθεί. Ε, ξέρουμε βεβαίως ότι ζούμε μια δύσκολη περίοδο στην Ευρώπη. Αν θέλουμε όμως ε, να προοδεύσουμε θα πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και την εκπαίδευση. Γιατί τότε θα έχουμε και κάτι να αποκομίσουμε από αυτή την επένδυση. Θα τα πάρουμε πίσω τα χρήματά μας εντός αγικών. Πάντα μπορούμε να κάνουμε περικοπές, αλλά η έρευνα είναι κάτι το οποίο μπορεί να διασφαλίσει την ανάπτυξη και την προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη. Και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε και να στηρίξουμε τέτοιου είδους προγράμματα. Σε γενικές γραμμές, αν τα κράτη-μέλη θέλουν να κάνουν περικοπές για τον έναν ή τον άλλον λόγο, εγώ ελπίζω να μην γίνουν περικοπές στην ανώτερη έρευνα. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε πραγματικά. Πρέπει να επενδύσουμε στο top research, στην, στα ανώτατα επίπεδα έρευνας και ίσως να γίνουν περικοπές στη βασική έρευνα. Αυτά είχα να πω. Βεβαίως ε, μπορώ να κάνω και άλλες παρατηρήσεις και άλλα σχόλια για τα όσα είπαν άλλοι συνάδελφοι για την καινοτομία και τις ανθρωπιστικές σπουδέ Θα πρέπει να υπάρχει πράγματι μια μεγαλύτερη ε, διασύνδεση μεταξύ των δύο. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε, αλλά συμφωνώ και με τα όσα είπε ο συνάδελφο κ. Σκέλη που μίλησε για τον αθλητισμό. κατά την αντιμετώπιση των ε, σύγχρονων προκλήσεων στις κοινωνίες μας. Και στην αρχή μίλησα για την σύνδεση μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης. Μια αντίστοιχη σύνδεση θα πρέπει να κάνουμε και μεταξύ έρευνας και αθλητισμού. Και αυτό είναι ένα ε, τομέα στον οποίο θα πρέπει να επενδύσουμε και μάλιστα στον αθλητισμό από μικρή ηλικία. Πράγματι, προσφάτως, πολλές ασθένειες που συνδέονται με την παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο και τα λοιπά, ε, έχουν αυξηθεί τα κρούσματα αυτών των ασθενειών. Αν λοιπόν επενδύσουμε περαιτέρω στην καινοτομία, στην έρευνα, την εκπαίδευση και τον αθλητισμό, τότε θα δημιουργήσουμε περισσότερη προστιθέμενη αξία. Όχι έρευνα για την έρευνα, λοιπόν. Έρευνα για ε, να, να ε, η κοινωνία. Γενικώ, Πρόεδρε, δεν ξέρω αν ε, κατάφερα να επιφέρω κάτι παραπάνω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά η κυρία Μακλάρκιν, όπως είπα και στην αρχή, βρίσκεται στο σωστό δρόμο και εγώ είμαι διατεθειμένος να στηρίξω ό,τι κάνει. Ελπίζω να έβαλα κι εγώ το λιθαράκι μου στο έργο της. Και πρέπει να είμαστε αυστηροί κατά τη συζήτηση αυτών των ζητημάτων στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Ρίβ. Φυσικά, εάν θεωρεί σκόπιμο να παρέμβει. thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία να λάβω το λόγο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την σημαντική της συμβολή στο θέμα αυτό. Όπως ξέρετε, η πρόταση Horizon 2020 έχει τρεις κυρίως στόχους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση που είναι μια πρόκληση για όλους. Δεύτερον, είναι μια ειλικρινής προσπάθεια να μετατοπίσουμε την έμφαση στα ερευνητικά θέματα με αυτούς που βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες της Ευρώπης. Το βλέπετε αυτό στο τμήμα που έχει να κάνει με τις κοινωνικές προκλήσεις και τρίτον, και αυτό είναι κάπως παστικό και ρηξικέλευτο, αν το συγκρίνετε με το πρόγραμμα πλαίσιο πριν από 10 χρόνια, βλέπετε πόσο μεγάλη αλλαγή έχει επέλθει. Το τρέχον αυτό, το επερχόμενο πρόγραμμα πλαίσιο, έχει βέβαια τον πυλώνα της επιστήμης που έχει σαν στόχο να ενισχύσει τη συνολική θέση της ε, ευρωπαϊκής ε, Ένωση την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Αναφέρθηκαν πάρα πολλά κατά τη διάρκεια τη συζήτησης. Ίσως δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλα τα στοιχεία, θα κάνω όμως κάποια σύντομα σχόλια για τα περισσότερα θέματα που ηγέτησε. Το στοιχείο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταρχήν τονίστηκε. Προφανώς και η πρότασή μας περιλαμβάνει μια σαφή και έντονη έμφαση για το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έχουμε και ένα ιδιαίτερο εργαλείο, ιδιαίτερο μέσο που προσπαθεί να δώσει συνέχεια στο γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο για την αγορά, οπότε πρέπει να έχουν έρευνα που να είναι πιο φιλική προς την αγορά. Έχουμε το στόχο 15% του προϋπολογισμού για τις κοινωνικές προκλήσεις και τις ε, ηγετικές τεχνολογίες να δαπανηθούν με πρόσθεση μάλλον τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υποστηρίζουμε το πρόγραμμα Eurostart, την καινοτομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά έχουμε και ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου. Με την πλατφόρμα ε, χρέους και μετοχικού κεφαλαίου. Όλα αυτά καταδεικνύουν το ότι υπάρχει μια μετακίνηση από την προηγούμενη εμπειρία του 7ου προγράμματος πλαισίου όπου υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως φάνηκε και από την έκθεση της κυρίας Έρικα Μάν που ήταν προηγουμένως <clears throat> βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το οποίο επίσης μας ενδιαφέρει είναι το να εξασφαλίσουμε μια ευρύτερη συμμετοχή, κάτι το οποίο έχει αναφερθεί πολλές φορές, να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι παρά το ότι όπως τονίζουμε συνέχεια και δεν το διαμφισβητεί κανείς, θα πρέπει να χρηματοδοτεί τις ενέργειες και τα προγράμματα αριστείας στο πρόγραμμα πλαίσιο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει και μια γενικότερη υποστήριξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό συμμετοχής κτλ. Και θα δείτε ότι υπάρχουν κάποια ειδικά μέτρα μέσα στο πλαίσιο της περιεκτικότητος για τις κοινωνικές προκλήσεις, για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού κτλ. που αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό του πώς θα μπορέσουμε να διευρύνουμε την συμμετοχή, <clears throat> παραδείγματο χάρη, με το να συνδέσουμε αναδυόμενα ιδρύματα, ε, κέντρα αριστείας και ιδιαίτερες περιφέρειες για να προσελκύσουμε ακαδημαϊκούς υψηλού επίπεδου και να συνεργαστούμε με ξένα ερευνητικά κέντρα. Όλα αυτά λοιπόν είναι και η απάντηση που δόθηκε στα θέματα αυτά μετά από σημαντική επεξεργασία που έλαβε χώρα πέρσι και πράγματι προέκυψε και από την ενδιάμεση αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαισίου. Τώρα για την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι λαθασμένο να πιστεύει κανείς ότι το ορίζον 2020 δεν θα χρηματοδοτήσει την πολιτιστική κληρονομιά. Οι προτάσεις μας είναι πάντα σύντομα <clears throat> έγγραφα που καλύπτουν ευρείες περιοχές χρηματοδότησης οι οποίες στη συνέχεια καθορίζονται πιο λεπτομεριακά. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο περιθώριο για χρηματοδότηση σχεδίων στον πολιτιστικό τομέα. Αυτό μπορεί να γίνει και από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο εξάλλου. Υπάρχει ιδιαίτερη μνήμα για τα πολιτιστικά θέματα στο κείμενο που καταδεικνύει και πώς η εφαρμοσμένη έρευνα μπορεί να χρηματοδοτηθεί <clears throat> και η ηγετική, η πρωτοποριακή έρευνα στη βιομηχανία. Σε διάφορα σημεία λοιπόν του κειμένου αναφέρεται η, ο τομέας της δημιουργίας όπου λέει ότι με τη χρήση συγκλουνσών τεχνολογιών μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες υπηρεσίες, νέες επιχειρήσεις που προστατεύουν και ενισχύουν την πολιτιστική αξία κτλ. Αναφέρεται επίσης ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας στην πρότασή μας για τον ορίζοντα 2020 και εν πάση περιπτώσει αυτό το... αυτή η πρόταση είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με το πλαίσιο της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένα στοιχεία του Horizon 2020, οι υποτροφίες Marie Curie, υποστήριξη για τους νέους, όλα αυτά είναι στοιχεία της οικοδόμησης ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού χώρου και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι και μέσα στο κείμενο αυτό υπάρχει έμφαση στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση και σε δράσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την κατανόησή μας της εξέλιξης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου. Τα προβλήματα της διάστασης του φύλου είναι κάτι το οποίο έχει αναφερθεί επίσης. Βλέπουμε σαν εγκάρσιο θέμα το φύλο για όλα αυτά τα προγράμματα του Horizon 2020. Πώς θα αντιμετωπιστούν λοιπόν τα θέματα ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών. Αυτό είναι βασική μέρημνα του προγράμματος. Και βέβαια κανείς δεν λέει ότι αυτό το πρόβλημα δεν υπήρχε στο παρελθόν και έχει επισημανθεί από προηγούμενες ε, αξιολογήσεις του έκτου προγράμματος πλαισίου και η διάμεση αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου και βλέπετε από την απάντηση που έδωσε η Κομισιόν και στα δύο αυτά έγγραφα το πόσο σημαντικό θεώρησε η Κομισιόν το να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Αναγνωρίζουμε ότι ένα τμήμα του προβλήματος είναι ο χαρακτήρας της επιστημονικής εργασιακής αγοράς στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά, η Κομισιόν το παίρνει πολύ στα σοβαρά. Και επίσης τα θέματα αυτά θα αντανακλώνται οι ισότητα των φύλων και στις συμφωνίες για χορηγήσεις. Το πρόγραμμα μας επίσης είναι ένα πρόγραμμα διεθνούς χαρακτήρα. 169 διαφορετικές χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα πλαίσιο, που είναι ένα εκπληκτικό επιτάγμα. Και η πρόταση Horizon 2020 θα εξακολουθήσει να τονίζει τη σημασία των διεθνών συνεργασιών. Με κάποιες αποχρώσεις θα υπάρξει κάποια μεγαλύτερη ε, εστίαση στη χρηματοδότηση, ώστε να βοηθηθούν και λιγότερο πλούσιες χώρες και θα υπάρχει και μεγαλύτερη έμφαση στην πρόσβαση στα προγράμματα αυτά. Μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε και εταιρικέ σχέσεις με τα κράτη-μέλη μέσω κοινοπραξιών με εταίρους από τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Ο προϋπολογισμός επίσης για το Horizon 2020 αναφέρθηκε. Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Κανείς δεν θεωρεί ότι οι συζητήσεις τους επόμενους μήνες θα είναι εύκολες. Το ποσό στο οποίο καταλήξαμε ήταν αποτέλεσμα μιας λεπτομερούς ανάλυσης από την Κομισιόν, αλλά η υποστήριξή σας, η, η θέλησή σας να αυξηθεί αυτό το ποσό είναι ιδιαίτερα καλόδεκτη. Αναφέρατε επίσης τη σημασία Τη σύνδεσης της έρευνας με την παιδεία. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, είναι εγγενές μέσα στην συνεργατική αυτή δράση του Horizon 2020 και ο αθλητισμός αναφέρεται πολλές φορές. Και κατανοώ αυτό που λέτε ότι ίσως το κείμενο θα μπορούσε να τονίζει περισσότερα τα θέματα του αθλητισμού. Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις όπου οι δραστηριότητες αυτές που αναφέρεται οι προκλήσεις για την υγεία, τα νέα υλικά, νανοτεχνολογία κτλ πάντα ο αθλητισμός θα είναι ένας χώρος όπου θα υπάρχει η έρευνα για νέα υλικά και νέες δραστηριότητες και επίσης η πρόκληση για την περιεκτικότητα θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πλειάδα ευρυτέρων πρόγραμμα προβλημάτων κοινωνικών που συνδέονται με τον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων Εάν μου επιτρέπετε και η συνάδελφός μου θα ήθελα να πει κάτι για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα... Μήπως μπορείτε να πείτε το όνομά σας παρακαλώ. Ruth Χάιτ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Παλιαδέλη για το ερώτημά της ε, για το Ίδρυμα EIT. Ε, για να διευκρινίσω, είναι σαφές ότι το Ίδρυμα αυτό είναι ένα ανεξάρτητο Ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου. Ο στόχος του είναι να συγκεντρώσει πόρους, όχι να δαπανίσει πόρους. Ε, ε, ε, αυτό ισχύει για το ένα. Εδώ είναι άλλος ο ρόλος του εδώ. Είναι να χρηματοδοτήσει δράσεις να, προσπαθήσει να ενοποιήσει το τρίγωνο της μάθησης. Υπάρχει επικέντρωση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το ε, Ίδρυμα έχει ξεκινήσει τις εργασίες του, το πρόγραμμα εργασίας του το υλοποιείται ήδη. Αλλά ε, για παράδειγμα, θα στηρίξει τους φοιτητές, θα στηρίξει το ταλέντο, την κατάρτιση. Ελπίζω έτσι να σας έχω ξεκαθαρίσει λίγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή και τώρα ο λόγος στην αγαπητή κυρία Μακλάρκεν, την εισηγήτρια, για να μας δώσει τα συμπεράσματα της συζήτησης. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τις συνεισφορές σας. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί ξέρω ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Αλλά το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ για τις συνεισφορές σας, για το πάθος σας, για τον οράζοντα 2020. Πραγματικά πολύ ωραία θέματα, γυναίκες και επιστήμη, η σύνδεση μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων που υλοποιούνται, η σύνδεση με το Εράσμους, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την έρευνα, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, θέλουμε να αναπτύξουμε γενικά την έρευνα ε, και γενικά να δούμε πού συνδέεται ο ένας τομέας και η μία θεματική με την άλλη. Επίσης πρέπει να παράγουμε αποτελέσματα. Και σας ευχαριστώ πολύ για την έμφαση στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Ε, που είπε η κυρία Σμιτ. Επίσης, ε, η προσβασιμότητα στους πόρους αυτούς πρέπει να είναι πολύ εύκολη, όσο το δυνατόν πιο εύκολη για όλους όσους θα ζητήσουν πόρους. Πρέπει πραγματικά να παρέχουμε και την περίφημη προστιθέμενη αξία. Αλλά προς την Επιτροπή και τους ε, συναδέλφους θέλω να επαναλάβω την προσήλωσή μου στο ζήτημα. να λαμβάνεται υπόψη η πολιτιστική διάσταση. Δεν θέλω αυτό να μένει στα μικρά γράμματα. Δεν θέλω να είναι ένα παρεπόμενο. Όχι. Επίσης, οι δημιουργικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού. Θέλω να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα σε αυτές. Αυτά ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Σας θυμίσω ότι και για τα δύο σχέδια χνομοδότησης, σημεία 4 και 5, αυτά θα παρουσιαστούν τον Μάιο και θα τα ψηφίσουμε τον Ιούλιο. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε αυτή τη μεγάλη αίθουσα γιατί θα έχουμε μια δημόσια ακρόαση για τον καθορισμό του, του μελλοντικού προγράμματος της Ευρώπης για την εκπαίδευση και την ε, νεότητα, την νεολαία. Και σας ε, παροτρύνω να συμμετέχετε. Και τώρα περνάμε στο σημείο 6 που αφορά πάντα μια γνωμοδότηση νομοθετική, ε, συναπόφαση πρόταση για μια οδηγία που τροποποιεί την οδηγία του 2003 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Ο γενικός στόχος αυτής της οδηγίας είναι να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο ε, στο πλαίσιο του οποίου οι δημόσιες αρχές διαθέτουν στο κοινό τις πληροφορίες που έχουν ε, και την απάλληψη της ε, αδιαφάνειας και της ε, μη δίκαιης ε, και ίσης πρόσβασης χρήσης των πληροφοριών αυτών σε όλους. Το κοινό θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση και να μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα όλες τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι δημόσιες αρχές. Προτάσεις για τη βελτίωση των βιβλιοθηκών, των δημόσιων αρχείων, κτλ. Η Επιτροπή Ήτρε, υπεύθυνη επί της ουσίας, θα υποβάλει το σχέδιο τον Ιούλιο και θα ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Σήμερα ε, ο εισηγητής μας, ο κύριος Φερχάιεν, θα μας εξηγήσει τα βασικά σημεία. Ε, το σχέδιο γνωμοδότησης θα παρουσιαστεί τον Μάιο, θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο και τώρα ο λόγος στον κύριο Φερχάιεν. Ähm, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί ήδη έχουν εφαρμοστεί πολλά στοιχεία της προηγούμενης οδηγίας. Εδώ υπάρξει μια βελτίωση του τρόπου υπολογισμού και της διεύρυνσης της εμβέλειας της οδηγίας. Πρόκειται για το πώς να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία στις βιβλιοθήκες, ακόμα και τις πανεπιστημιακές, στα αρχεία και στα μουσεία. Καταρχήν αυτό είχε δημιουργήσει κάποια ανησυχία, αλλά δεν θα εφαρμοστεί στα ερευνητικά ιδρύματα αυτά κάθε αυτά ή σε καλλιτεχνικούς οργανισμούς όπως είναι μπαλέτα, θέατρα κτλ. Θα περιοριστεί μονάχα σε βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία. Τώρα η περαιτέρω διεύρυνση στα ραδιόφωνα, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς δεν είναι κάτι το οποίο προβλέπεται σε αυτή την οδηγία. Αποκλείονται προς το παρόν όλα αυτά. Η επέκταση αυτή του πεδίου εφαρμογής ε, περιορίζεται μονάχα στις βιβλιοθήκες, στα αρχεία και τα μουσεία, γιατί αλλιώς υπάρχουν πολλά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν για την ερευνητική δραστηριότητα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν παραδείγματος χάρη προβλήματα συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων και γι' αυτό το λόγο είναι λογικό πιστεύω να υπάρξει αυτή η εξαίρεση των τομέων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να αναμείνουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε περισσότερη διεύρυνση της εμβέλειας της οδηγίας. Ε, είναι σημαντικό επίσης και για τα ραδιόφωνα να βρεθούν εκτός αυτής της ε, οδηγίας γιατί πολλές φορές βασίζονται σε οι εκπομπές σε λεγόμενα ορφανά έργα και πρέπει επομένως να αποκλειστούν στοιχεία τα οποία έχουν copyright, υπόκειται ακόμα σε copyright και δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε αυτή την ενέργεια σε σχέση με το κόστος το οποίο θα προέκυπτε. Γιατί το κόστος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο βάσει της πρότασης Κομισιόν τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων θα μπορούν να συλλέγονται από τους οργανισμούς αυτούς, αλλά επίσης και με την αναπαραγωγή, ε, θα, μάλλον θα περιορίζονται στο κόστος αναπαραγωγής αυτών των έργων. Ο στόχος είναι λοιπόν να υπάρξουν τέτοιου είδους περιορισμοί για τα τέλη τα οποία μπορούν να προκύψουν. Εγώ θεωρώ ότι είναι θετικό αυτό ως ρύθμιση από τη μία πλευρά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το κόστος το οποίο προκύπτει στην πραγματικότητα από την ε, έκδοση και την ε, διαθεσιμότητα σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Ο στόχος μας είναι να μην υπάρξουν πρόσθετα κόστη, κόστη που έχουν να κάνουν με τη χρήση προσωπικού και τα οποία να μετακυλιστούν στον χρήστη αυτών των υπηρεσιών η Κομισιόν θα πρέπει να ελέγξει ακόμα περισσότερο σε επίπεδο έκθεσης αντικτύπου ποιες μορφές ε, κόστους προκύπτουν από την χρήση ηλεκτρονικής μορφής για αυτά τα έγγραφα και επίσης για την χρήση ε, μορφής των εγγράφων αυτών που να είναι αναγνώσιμα από υπολογιστές. Τίθεται εδώ το ερώτημα του αν υπάρχει μονάχα ένας δυνητικός αναχρησιμοποιητής αυτών των δεδομένων και δεν υπάρχει καμία περαιτέρω δυνητική χρήση αυτών των εγγράφων, με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να υπολογίσει το πρόσθετο κόστος επί τη βάση της ζήτησης αυτών των, ε, του ενός μονάχα χρήστη. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να είναι υπολογίσιμη και διερευνήσιμη η πηγή κάθε περιττέρω κόστους ώστε να μην καταλήξουμε σε μια υπερβολικά περιοριστική ε, ρήτρα στην οδηγία αυτή. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ιδίως για τα αρχεία και τα μουσεία και το οποίο παίζει πάντα ρόλο και στο, και στο σχέδιο Ερωπεάνα είναι η υποστήριξη προς ε, ε, υπηρεσίες που δεν έχουν τα κονδύλια να μπορέσουν να προχωρήσουν σε ψηφιοποίηση βιβλίων, πινάκων ε, κτλ. Και θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη για να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικούς εταίρους σε αυτή τη δραστηριότητα, αλλά αυτό μονάχα μπορεί να γίνει εάν υπάρξει μια αποκλειστικότητα από αυτή την άποψη. Αλλιώ οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς δεν νομίζω θα δείξουν ενδιαφέρον. Έτσι τα μουσεία και τα αρχεία μπορούν να έχουν μια αποκλειστική συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς προς τον στόχο της ψηφιοποίησης και της επίτευξης προσθέμενης αξίας στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιτρέπεται να έχουμε μια τέτοια δραστηριότητα. Διαλειτουργικότητα τώρα. Η πρόταση της Κομισιόν λέει τώρα ότι θα πρέπει να απλοποιηθεί η λειτουργία με την δημιουργία ενός κοινού πλαισίου μηχανικά αναγνώσιμων εγγράφων που θα εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα. Εδώ θα προτιμούσα μια καλύτερη διατύπωση η οποία θα εξασφαλίσει ότι δεν υποχρεωμένοι όλοι να χρησιμοποιούν έγγραφα σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή μονάχα, γιατί αυτό προϋποθέτει και πρόσθετο κόστος. Αρκεί να είναι σε, στα συνηθισμένα φόρμα αυτά τα έγγραφα, επί τη βάση των οποίων μπορεί κανείς να τα μετατρέψει σε μια μορφή η οποία είναι προσβάσιμη και στους αναγνώστες αλλά και σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν την αναλογικότητα όλων αυτών των μέτρων και να μην είμαστε υπερβολικοί. Κάτι ακόμα το οποίο αντιμετωπίζω στην έκθεσή μου είναι το θέμα των ανεξαρτήτων αρχών όπως προτείνει η Κομισιόν. Λέει η Κομισιόν ότι αυτός ο οποίος κάνει μια αίτηση εάν υπάρξει μια άρνηση στην πρόσβαση θα πρέπει να έχει την δυνατότητα πρόσβασης και προσφυγή σε μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα κάνει τον έλεγχο των αποφάσεων των αρχών που έχουν να κάνουν πρόσβαση σε αυτά τα δημόσια έγγραφα. Η πρόταση μιας ανεξάρτητης αρχής για μένα σημαίνει περισσότερες γραφειοκρατικές δομές και το να έχουμε ακόμα περισσότερο συγγνώμη. Μήπως μπορείτε να τα λέτε λίγο πιο αργά, μήπως τα καταφέρουν και σας παρακολουθήσουν και οι διερμηνείς, λέει ο πρόεδρος. Αν λοιπόν κάθε κράτος μέλος υποχρεωθεί να έχει τη δικιά του ανεξάρτητη αρχή για τα θέματα αυτά, αυτό θα οδηγήσει σε ένα δυσανάλογο κόστος και στην ανάγκη δημιουργίας προσθέτων εποπτικών αρχών. Θα είχε νόημα λοιπόν αυτό αν έχουμε μία δομή που ως μορφή κοιτίου παραπώνου θα μπορούσε να λειτουργεί. Αλλά μια ανεξάρτητη αρχή για μένα είναι κάτι το υπερβολικό. Είναι ασαφής λοιπόν η πρόταση κομισιών πού θα βρίσκεται αυτή η ανεξάρτητη υπηρεσία και πώς θα έχει αντιμετωπιστεί από κάθε κράτος μέλος, δεν ξέρω και αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως έχει να κάνει με την αρχή της επικορικότητας κάθε κράτος μέλος, έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αφ' αυτού τι θα κάνει με αυτή την αρχή και δεν θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται ως ξεχωριστές κεντρικές αρχές. Εν γέννη λοιπόν μπορούμε να χαιρετήσουμε αυτή την πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας και νομίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος μας για την τροποποίηση αυτή να μην προκύψει δυσανάλογο κόστος το οποίο δεν έχει καμία αξία και να μπορούμε να έχουμε την σωστή χρηματοδότηση στο επίπεδο που χρειάζονται αυτές οι υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος, η κυρία Κάμερβερτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ζαμπίνε. Νομίζω ότι δεν έχουμε μεγάλες διαφορές σε σχέση με την έκθεση αυτή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία εγώ θα ήθελα να θέσω για την οδηγία αυτή. Ιδιαίτερα το άρθρο 6 το οποίο μου φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα. Λέμε από τη μια μεριά ότι δεν πρέπει να υπάρξει κάποιο κέρδος από τις δραστηριότητε αυτές. Αυτό είναι φυσιολογικό <clears throat> για το δημόσιο τομέα. Από την άλλη μεριά λέμε ότι κάθε μορφή κόστους η οποία θα προκύψει θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα τέλη. Και όπως το έχει διατυπώσει λοιπόν η Κομισιόν, δεν είναι ιδιαίτερα σαφές αυτό. Μήπως θα ήταν καλύτερα να σκεφτούμε αν τα μουσεία, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ε, θα μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετα τέλη, αλλά να αναφέρεται ακριβώς πού βρίσκονται αυτά τα τέλη. Αλλιώς εμείς κάνουμε μια, έχουμε μια διαφορετική μεταχείριση των αρχείων, των βιβλιοθηκών και των μουσείων και άλλων δημοσίων φορέων που μπορούν να επιβάλλουν μόνο περιορισμένα τέλη για να καλύψουν το κόστος τους. Θα πρέπει να είναι εκπεφρασμένο ποια είναι αυτά τα στοιχεία κόστους τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και εγώ βλέπω να είναι προβληματικό να δημιουργήσουμε μια πρόσθετη ανεξάρτητη αρχή. Δεν ξέρω τι ακριβώς προβλέπει η Κομισιόν, τι στοχεύει να κάνει η Κομισιόν, είναι μια δομή σε κρατικό επίπεδο, σε κάθε κράτος μέλος ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ υπάρχει και το θέμα της ισότητας ανταγωνισμού και της προστασίας στοιχείων. Μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση που θα υπάρχουν προβλήματα αν κάθε φορά δημιουργούμε τέτοιους φορείς που θα επικαλύπτονται οι αρμοδιότητες τους με άλλων φορέων. Θα πρέπει εδώ λοιπόν να έχουμε την απαραίτητη διευκρίνηση. Επομένως υποστηρίζω σε γενικές γραμμές όλα αυτά που είπε η Σαμπίνε και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε αρκετά σύντομα να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση σε σχέση με τη γνωμοδότησή μας για την τροποποίηση αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο Σαμπίν Παγάιεν. Ίσως λόγω της ταχύτητας Άκουσα πολλά για το κόστος και όχι και πολλά για τα ωφέλη. Ποια είναι λοιπόν τα ωφέλη για αυτά τα ανοιχτά δεδομένα στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Εδώ μπορούμε να είμαστε και φιλόδοξοι και για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για την θέση της Ευρώπης στον κόσμο, γιατί δεν εξετάζουμε μόνο εμείς αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Είναι σημαντικό η Επιτροπή εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει τον δεχόμενο συμπερίληψη περισσότερων ε, ε, πληροφοριών στην αναθεωρημένη οδηγία. Γιατί όταν αυτά χρηματοδοτούνται ήδη από τα δημόσια κονδύλια, ήδη οι πολίτες έχουν πληρώσει ένα μεγάλο μέρος αυτής της διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές ε, διαφωνίες αυτή τη στιγμή και είναι σημαντικό να δούμε πώς εξετάζουμε την έννοια του κόστους και την έννοια του ωφέλους. Ας εξετάσουμε τη διαφωνία μεταξύ των ε, ακαδημαϊκών ερευνητών και των εκδοτικών οίκων. Πολλοί ε, εκδότες θεωρούν ότι έχουν τα πνευματικά δικαιώματα για, τους, για, το αποτέλεσμα των ερευνών και πολλούν εκ νέου τις έρευνες ε, στα πανεπιστήμια. Και τα πανεπιστήμια πρέπει να πληρώσουν δεκάδε χιλιάδε ευρώ ε, για, σε πνευματικά δικαιώματα για να βρουν το, το δικό του αρχικό έργο. Επομένως, ε, το κοινό πληρώνει για την ε, ε, δημιουργία νέας επιστημονικής γνώσης και ξαναπληρώνει για την ίδια γνώση στους εκδότες. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να ε, συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε μια πιο συνδεδεμένη, αν θέλετε, ψηφιακή κοινωνία. Υπάρχουν πολλές βέλτιστες πρακτικές σε, σε κορυφαία επιστημονικά Ινστιτούτα στον κόσμο όπως το MIT που έχει ανοίξει ε, την πρόσβαση στο επιστημονικό του υλικό και δίνει πρόσβαση σε τέτοιο υλικό σε δεκάδες χιλιάδες ε, ε, πολίτες. Υπάρχει και το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης και εκεί είναι σημαντικό να δούμε πώς η ανταλλαγή επιστημονικών επιστημονική ε, γνώση μπορεί να οδηγήσει σε ωφέλη. Αυτό ισχύει για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο του Ντέλφτ, ε, που είναι πρωτοπόρο σε ό,τι αφορά την διαχείριση υδάτων. Και ε, πολλέ από, το, το, αποτέλεσμα της γνώσης που παράγεται εφαρμόζεται σε πολλές χώρες όπως ο χώρες της Αφρικής και εκεί βλέπουμε και την πρακτική εφαρμογή του επιστημονικού υλικού. Στην πράξη δηλαδή αντεκατοπτρίζεται ε, και υλοποιείται στην πράξη κάτι το, στην Αφρική κάτι το οποίο έχει παραχθεί στις ε, κάτω χώρες. Αυτό μπορεί να ισχύσει και για, τις, ε, για την πολιτιστική κληρονομιά, την πολιτιστική παραγωγή και η Σαμπίνα αναφέρθηκε σε πολλά τέτοια σημεία. Έχουμε τέτοια πολυμορφία στον πολιτισμό και τέτοιο πλούτο που αποκρύπτουμε προς το παρόν από το κοινό. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ανοιχτή πρόσβαση σε όσους τον περισσότερους πολίτες. Και για το τι μπορεί, πώς μπορεί να αξιοποιήσει ο κόσμος αυτά τα στοιχεία, αυτό δεν είναι εύκολο να το προβλέψουμε. Πώς δηλαδή το κοινό θα αξιοποιήσει τις ε, διαθέσιμες πληροφορίες. Όμως ε, εκπήρα σε άλλους τομείς, για παράδειγμα στις ε, πληροφορίες για τον καιρό ή για τις μεταφορές, είδαμε και στοιχεία καινοτομίε από, τον κοινό, από το κοινό. Οι προγραμματιστές, για παράδειγμα, δημιούργησαν ένα σύστημα μεταφορών, ε, πληροφόρησης για τις μεταφορές σε πραγματικό χρόνο. Οι πολίτες δηλαδή ξέρουν πότε ακριβώς θα φτάσει το λεωφορείο, όχι μόνο τι λέει το χρονοδιάγραμμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τι γίνεται με τι βέλτιε πρακτικέ. Ε, σε κάποια κρατημέλη, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο και οι κάτω χώρε, έχουν ηγετικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα και συμφωνώ με τα όσα είπαν οι άλλοι συνάδελφοι. Να μην υπάρχει κανένα επίπεδο γραφειοκρατία. Να αφαιρέσουμε από την γραφειοκρατία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καβαδά. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για το μέγεθος ουσιαστικά και τον πλούτο αυτού του φακέλου. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία μονάχα. Δεν πιστεύω ότι αν υπάρχει μια σύγκρουση, μια διαμάχη, θα είναι καλή ιδέα να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αρχή. Πρώτα απ' όλα τα κράτη-μέλη έχουν σχεδόν όλα τις ε, εθνικές αρχές, οι οποίες λειτουργούν λίγο πολύ καλά όσο φυσικά τα κράτη-μέλη, οι κυβερνήσεις κρατάνε μια απόσταση ασφαλείας από όλα αυτά τα θέματα, κάτι το οποίο δεν γίνεται πάντα. Όταν υπάρχει πάντα λοιπόν μια και όταν καταλήγουν τα πράγματα σε ανοιχτή διαμάχη θα πρέπει να καταλήξουν στα δικαστήρια. Πιστεύω μια Ευρωπαϊκή Αρχή θα κατέληγε σε μια ιδιαίτερα γραφειοκρατική αντιμετώπιση όπως και σε πολλούς άλλους τομείς έχουμε δει. Επομένως αυτή την ιδέα θα πρέπει να την απορρίψουμε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, εάν επιθυμεί να προσθέσει κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω το όνομά σας, έχω κάποιο πρόβλημα, αλλά αν θέλετε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Λέγομαι Σουέτεναν. Είμαι επικεφαλής της μονάδος για την ε, πρόσβαση ε, στην πληροφορία και τη γενική, στη Γενική Διεύθυνση για την Πληροφορία και τα Μέσα Ενημέρωσης. Εγώ άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον όλα τα σχόλια των ε, μελών σήμερα είναι σαφές ότι πολλά από τα ζητήματα τα οποία έχουν αγερθεί από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου μπορούν να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη, ε, με μεγαλύτερη διαλεύκανση, αν θέλετε, των προτάσεων της Κομισιόν. Γιατί η πρότασή μας ίσως δεν ήταν τόσο σαφής όσο θα θέλαμε να είναι, παρόλα αυτά. Η διαδικασία, η νομοθετική στην οποία συμμετέχουμε με τις δύο νομοθετικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω θα βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε λίγο καλύτερα όλα αυτά τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν από την κυρία Φερχάιεν και για τα οποία έχουν αναφερθεί και άλλοι ομιλητές. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω τώρα τις ευρύτερες πλευρές που ανέφερε και η κυρία Σάκε. Εδώ η πρόταση της Κομισιόν είναι τμήμα ενός ανοιχτού πακέτου που συνοδεύεται από μία ανακοίνωση της Κομισιόν και η Κομισιόν είναι το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο έχει εγκρίνει μία απόφαση αυτού του είδους. Πιστεύω ότι αυτό, αυτή η ανακοίνωση ενθαρρύνει και τα άλλα θεσμικά όργανα να προχωρήσουν προς την ίδια κατεύθυνση και υπάρχει αυτή η κατεύθυνση ανοιχτών δεδομένων που για λόγους και διαφάνειας και για λόγους οικονομικούς θέλει να παροτρύνει όλους να κάνουν μια καλύτερη χρήση των πληροφοριών που έχουν συλλεγεί από δημόσιους φορείς ως τμήμα των αρμοδιοτήτων τους και που μπορούν στη συνέχεια αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν και για άλλους στόχους. Το θέμα της καταβολής τελών είναι προφανώς ένα από τα κεντρικά ζητήματα τα οποία γύρονται. Η μελέτη μας για τα θέματα αυτά κατέδειξε ότι το να επιβάλλουμε τέλη παρά το γεγονός ότι οδηγεί σε κάποια συλλογή ε, χρημάτων συμπεριλαμβάνει και κάποιο κόστος και τελικά είναι κάτι το αντιπαραγωγικό. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να περιορίσουμε το κόστος μονάχα στο οριακό κόστος και θέλουμε να περιορίσουμε την προσπάθεια των κρατών μελών και τον οργανισμό τους να ζητούν να συλλέξουν χρήματα από την επαναχρησιμοποίηση των εγγράφων αυτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε σε περισσότερη λεπτομέρεια όσο προχωρούμε στην νομοθετική διαδικασία, ώστε έτσι να καταλήξουμε στους νέους κανόνες οι οποίοι πρέπει να είναι πρόσφοροι και ορθοί. Θέλω να υπογραμμίσω ότι σε κανένα βαθμό, σε κανένα σημείο μάλλον η Κομισιόν δεν θέλει να δημιουργήσει μια νέα ευρωπαϊκή αρχή, ούτε να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν αυτά νέε αρχές για το σκοπό αυτό. Αλλά αυτό το έργο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από μια ήδη υπάρχουσα αρχή στα κρατημέλη. Ευχαριστώ. Κυρία Φερχάιεν, έχετε πάλι το λόγο αν θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία αναφέρατε. Θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω τις ε, Προτάσει και τα σχόλια των βουλευτών στο κείμενο τη γνωμοδότησής μου. Θα έχω την επόμενη εβδομάδα επαφέ με του κοιόδης συζητητέ. Σε ένα σημείο θέλω να σταθώ. Άκουσα ότι η Κομισιόν έχει δημιουργήσει ένα κατάλογο ερωτήσεων και απαντήσεων για το θέμα αυτό. Θα ήταν χρήσιμο να το έχει και η Επιτροπή μας αυτόν τον κατάλογο, γιατί σε ορισμένε περιπτώσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη σαφήνεια. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε ένα σημείο να πω ότι η γερμανική, αγγλική και γαλλική γλωσσική έκδοση δεν ήταν, τις οδηγίες αυτής δεν ήταν πάντα σύμμορφες σε σχέση με το περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασάφειες και προβλήματα. Θα ήθελα να ζητήσω από τις υπηρεσίες μετάφρασης να ξανακοιτάξουν τα θέματα αυτά και να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ αυτών των ε, γλωσσικών μορφών. Γιατί υπάρχουν δύο-τρία προβλήματα τα οποία επεσήμενα σε γλωσσικό επίπεδο είναι χρήσιμο σε αυτές τις τρεις τουλάχιστον βασικές γλώσσες να είναι ακριβώς το ίδιο το οποίο λένε τα κείμενα και να μην προκύψουν διαφορές από τα κείμενα. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε πολύ γρήγορα σε συμφωνία σε μερικά βασικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την χρήση ερευνητικών στοιχείων και σε ό,τι αφορά το θέμα του κόστους. Εγώ νομίζω ότι η Κομισιόν έχει αντιμετωπίσει μια πολύ σωστά, με πολύ σωστό τρόπο αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει να κάνει την επαναχρησιμοποίηση ελκυστική. Από την άλλη πλευρά βέβαια δεν πρέπει να υπάρξει πρόσθετο κόστος για τους δημόσιους οργανισμούς. Αυτός δεν είναι ο καλύτερος τρόπος χρησιμοποίησης των δημοσίων α, κονδυλίων και να μην ε, ουσιαστικά καλύπτει το κόστος το κράτος για ενέργειες που γίνονται από ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι στη συνέχεια ενθυλακώνουν την προσθέμενη αξία. Θα πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια σωστή ισορροπία στα θέματα αυτά. Νομίζω ότι έχουμε κάνει λοιπόν μια σωστή διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στην κυρία Σάκερ νομίζω ότι δεν πρέπει να κρύψουμε τα θετικά στοιχεία. Υπάρχει μια μεγάλη πρόοδος η οποία μπορεί να προκύψει από αυτήν την ε, ενέργεια και είναι χρήσιμο να μπορούν τα πανεπιστήμια να έχουν την ε, δημοσίευση των προϊόντων. Ούτως ή άλλως τα πανεπιστήμια τα οποία είναι <clears throat> δημόσια μπορούν πάντα να το κάνουν. Αν τώρα ένα πανεπιστήμιο χρειάζεται πρόσθετα κονδύλια και χρηματοδότηση, είναι φανερό ότι ο ιδιωτικός οργανισμός που δίνει τη χρηματοδότηση θα διεκδικήσει και ε, αποκλειστικότητα στη δημοσίευση αυτών των προϊόντων. Και όταν υπάρχει μια υποχρέωση να δημοσιεύει κανείς μόνο σε ορισμένα περιοδικά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Δεν πρέπει λοιπόν αυτά τα οποία προτείνουμε εδώ να θεωρηθούν ότι είναι ε, υποχρεώσεις, μπορούν πάντα να οδηγήσουν σε μια παρότρινση ώστε τα ερευνητικά αποτελέσματα όλο και περισσότερο γίνονται προσβάσιμα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν επειδή υπάρχει το γλωσσικό πρόβλημα το οποίο ανέφερε η κυρία Φερχάιν, να ρωτήσω σε ποια γλώσσα είχε δημοσιευτεί, είχε διατυπωθεί το αρχικό κείμενο. Δυστυχώ, ακούσαμε αυτά τα αρνητικά σχόλια από την εισηγήτρια. Θα έρθουμε σε επαφή με την υπηρεσία μας για να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα και να βρούμε μια λύση αν υπάρχει πράγματι διαφορά μεταξύ των ε, διαφόρων γλωσσικών εκδοχών. Επίσης, ε, θα μεριμνήσουμε το ώστε να διαμοιραστούν τα non-papers που έχουμε καταρτήσει σε όλες τις επιτροπές ε, που εξετάζουμε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Θέλω να υπενθυμίσω τώρα ότι το σχέδιο αυτογνωμοδότησης θα αντιμετωπιστεί τον, ε, θα εξεταστεί πάλι τον Μάιο και θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο. Περνάμε τώρα στο σημείο 5. Τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας αφορά στην περίπτωσή μας τη σχέση με εταίρους στο ανατολικό και νότιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρχουν στενότερες σχέσεις με τις χώρες αυτές και καλύτερη κινητικότητα και πιο έντονες επαφές στον τομέα της παιδείας, ιδίως μέσω του προγράμματος Έρασμος για όλους. Γι' αυτό εμείς συντάσσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Έχουμε πολύ στενά χρονικά περιθώρια, διότι η Επιτροπή ΑΦΕΤ, η Εξωτερικών Υποθέσεων που είναι αρμόδια από της θα ψηφίσει τον Ιούνιο. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Μάτουλα. Θα παρουσιάσει την πρότασή του τον Απρίλιο και θα ψηφίσουμε το Μάιο. Επειδή λοιπόν έχουμε αυτό το πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για την παρουσίαση των τροπολογιών στην, οδηγή, στην γνωμοδότηση αυτή, μετά από συμφωνία με τη Γραμματεία, προτείνω μόλις λάβετε το σχέδιο έκθεσης να υποβάλλετε και τις τροπολογίες σας. Ο κύριος Μάτουλα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, είπατε όσα ήταν απαραίτητα. Εγώ ήθελα να πω μόνο ότι το Ευρωπαϊκό ε, Μέσο Εταιρικών Σχέσεων για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας ε, είναι το μέσο που αξιοποιούν και τα 16 μέλη στην ε, Μεσογειακή Περιφέρεια και στον τομέα της ε, ανατολικής θερικής σχέσης. Και η Ρωσία συμμετέχει ως προς αυτό ε, για τους τομείς ε, της ενίσχυσης της διακυβέρνησης, οικονομικής ανάπτυξης, διασυνοριακής συνεργασίας και συμμόρφωσης των χωρών που αξιοποιούν αυτό το μέσο. Τη συμμόρφωσή τους λοιπόν ως προς τις ευρωπαϊκές αρχές για τη δημιουργία ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα πρόταση αφορά την γειτονία σε ένα νέο πολιτικό ε, πλαίσιο και βασίζεται σε συγκεκριμένους ε, στόχους που μειώθηκαν από 29 σε 6. Έχουμε και μια νέα αρχή της αμοιβαίας ευθύνης που επιτρέπει τη διαφοροποίηση μεταξύ των ε, εταίρων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει και το ε, αξιοκρατικό κριτήριο. Τα κονδύλια χρηματοδότηση θα είναι περίπου 18 δις για τα έτη 2014-2020 σε σύγκριση με τα 11 δις στον προηγούμενο προπολογισμό μέλος χρηματοδότησης θα καλύπτεται από το πρόγραμμα Εράσμους για όλους ε, με δύο ετήσιες κατανομές για τρία και τέσσερα χρόνια. Πολιτισμός, έρευνα, καινοτομία είναι τομείς που μπορεί να υπάρξει ε, βελτίωση Ε, μεταξύ της εγχώρια πολιτικής και του μέσου καλής γειτονίας. Ε, το ίδιο το κείμενο είναι αρκετά τεχνικό και συνδέεται με τον τρόπο κατανομής των κονδυλίων. Για την... Ε, προκειμένου να έχουμε περισσότερες πιθανότητε έγκρισης των τροπολογιών μα από την Επιτροπή ΑΦΕΤ, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, προτείνω τροπολογίε που συμπεριλαμβάνονται στον τομέα αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Εγώ συναντήθηκα με τους κοιόδης συζητητές, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και έχουμε συμφωνήσει επί της αρχής σε αυτό το θέμα. Από πλευράς μου, εγώ θέλω να συμπεριλάβω τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στους συγκεκριμένους ε, στόχους ε, του μέσου γειτονίας. Ε, ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα ήταν καλό να διατηρήσουμε τη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση σε περίπτωση που η Ευρώπη αποφασίσει να θέσει ένα τέλος ε, στις συνδέσεις της με συγκεκριμένα καθεστώτα. Γιατί αυτός ο τρόπος κατανομής των κονδυλίων μας επιτρέπει να διατηρούμε σχέσεις και δεσμούς ε, με την κοινωνία των πολιτών σε διάφορες χώρες με την αξιοποίηση της πολιτιστικής διπλωματίας. Εγώ ε, περιμένω τις ε, προτάσει σα για να τι περιλάβω στην έκθεσή μου. Η καταληκτική μερομηνία για την υποβολή τροπολογιών είναι πολύ κοντά, όπω αναφέρατε κι εσείς γιατί η αρμόδια επιτροπή θέλει να ψηφιστεί πολύ γρήγορα. Κύριος Μενέντες Δεβάγε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν φυσικά θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, καλή του διάθεση και την συνεργασία σε σχέση με την ε, γνωμοδότηση αυτή και όπως είπε και ο Πρόεδρος, επειδή είναι πολύ στενές οι χρονικές προθεσμίες, χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό. Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία της κουλτούρας ως παράγοντα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται μονάχα για την εμπορική μας ικανότητα ή τη στρατιωτική μας ικανότητα, αλλά και για την πολιτιστική μας πολυπικιλία που αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα. Η ικανότητά μας να επηρεάσουμε τον κόσμο και να διγίνουμε ελκυστικοί για τρίτες χώρες θα υποσκαφθεί εάν δεν έχουμε μια σωστή παρουσίαση των πολιτιστικών μας επιτευγμάτων. Μέσα στα πλαίσια της τωρινής έκθεσης το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι αντιμετωπίζουμε τους πιο κοντινούς μας γείτονες. Σε σχέση λοιπόν με το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης θα ήθελα να κάνω μερικές σύντομες σκέψεις οι οποίες νομίζω ότι μπορούν να είναι και η βάση των τροπολογιών που θα παρουσιάσω στο μέλλον. Από τη μία πλευρά θέλω για τους λόγους που ανέφερα να επιστήσω την προσοχή σας στο άρθρο 2 της προτάσεως της Κομισιόν ότι δεν αναφέρεται εκεί ο πολιτισμός σαν ένας από τους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής υποστήριξης. Θεωρώ ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πολιτιστικός παράγοντας. Και επομένως το άρθρο 2 της πρότασης θα πρέπει να αναφέρει και τον πολιτισμό και όχι όπως τώρα να τον αφήνει απ' έξω. Επίσης, νομίζω ότι η ανταλλαγή πολιτιστικών αξιών και η έκφραση της πολιτιστικής μας πολυμορφίας θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα και να περιλαμβάνεται στο άρθρο αυτό. Εξάλλου, βλέπω με ικανοποίηση ότι από ό,τι φαίνεται, λέω από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, το άρθρο 18.3 για το πρόγραμμα Έρασμος για όλους αναφέρεται ότι τα κονδύλια για το μέσο αυτό ε, συνεργασίας δεν θα προέρχονται από τα κονδύλια της Κομισιόν για αυτό το τομέα, αλλά από την, τον προπολογισμό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα μου φαινόταν επίσης πάρα πολύ χρήσιμο να ζητήσουμε από τις χώρες οι οποίες θέλουν να υποστηριχθούν από αυτό το εργαλείο να υποστηρίξουν τη σύμβαση της UNESCO για τη διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Σάντζε Σμιτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επιμείνω και πάλι σε μια πτυχή που αφορά την ε, περιφερειακή πολιτική στην παρουσίαση μιλήσαμε για τη διασυνεραϊκή συνεργασία σε αυτό το μέσο πολιτικής γειτονίας. Κάτι το οποίο μου φαίνεται ε, ένα μάλλον άγνωστο μέσο επιτρέπει την συνεργασία μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών ή των ε, περιφερειακών αρχών και επιτρέπει την διατήρηση σχέσεων ακόμα και αν υπάρξει ρήξη στις σχέσεις των ε, κρατών ε, ενέργειες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Επιτρέπει λοιπόν αυτό στην κοινωνία των πολιτών ε, των δύο χωρών να συνεργαστούν και να διατηρηθούν σχέσεις εκεί που υπάρχουν δυσκολίες μεταξύ των χωρών αυτών. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της ε, Επιτροπής θέλει να προσθέσει κάτι. Η Γενική Διεύθυνση για τη Διεύρυνση. Δεν υπάρχει κανείς. Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξωτερικών Σχέσεων ε, δεν υπάρχει, δεν είναι στην αίθουσα. Εντάξει, λοιπόν, ο λόγος ε, στον κύριο Μάντουλα για να προσθέσει κάτι και εκείνος. Foarte scurt, aș dori doar să mulțumesc colegilor și Πολύ σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τον κύριο Δεβάγε και την συνάδελφο Σάντσε Σμιτ για την στήριξη που έδειξαν στο πρόσωπό μου και για σε ό,τι αφορά την έκθεσή μου, αλλά και στην συμπερίληψη του πολιτισμού, της πολιτιστικής πτυχής, όπου ανήκει, για τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν, βεβαίω και για την Σύμβαση UNESCO. Ε, βεβαίω ε, είναι απολύτω ε, φυσικό και ελπίζω να συμβεί στο μέλλον. Η κυρία Σάντσε Σμιθ φυσικά και πολιτιστική διπλωματία πρέπει να είναι το κύριο μέσο που θα πρέπει να δημιουργήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και τη διατήρηση των εξωτερικών μας σχέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένω τις απόψεις σας ε, και ελπίζω να συνεργαστούμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Μάτουλα. Σας θυμίσω ότι ο συνάδελφος θα υποβάλει το σχέδιο τον Απρίλιο και θα ψηφίσουμε τον Μάιο. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης που είναι η online διανομή οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγητής ε, Καβαντά. Έχουμε κάνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων τον Ιανουάριο. Ε, θα παρουσιαστεί τώρα το σχέδιο του κειμένου. 12 ε, Απριλίου είναι η προθεσμία στις 12 η ώρα για την υποβολή τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο. Το λόγο έχει ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι η δημιουργική έκφραση των δημιουργών στον οπτικοακουστικό τομέα, στον κινηματογραφικό τομέα δεν είναι απλή υπόθεση γιατί εξαρτάται ε, ταυτόχρονα από την τέχνη αλλά και την οικονομία. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ευκαιρίες καθώς και μέσα διάδοσης των ευρωπαϊκών έργων γιατί η Ένωση θα πρέπει να προσανατολιστεί έντονα προς την παιδεία και τον πολιτισμό. Όπως πολύ συχνά λέγεται σε αυτή την αίθουσα, η δημιουργική και βιομηχανική κλάδη ε, αυτού του τομέα αντιπροσωπεύουν μεγάλη πηγή θέσεων εργασίας και η οικονομική συνεισφορά τους και η προστιθέμενη αξία τους υπολογίζεται στα 2,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ ε, σχεδόν το ίδιο με τα έσοδα από την αυτοκινητοβιομηχανία. Ε, θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο στο οποίο βασίζονται η εμπορία και διακίνηση ε, οπτικοακουστικών έργων ε, υπάρχει μια θηρίδα ειδικής εκμετάλλευσης εδώ, η οποία αντιστοιχεί στα διάφορα μέσα. Αυτό το σύστημα δεν πρέπει να το αμφισβητήσουμε όπως ισχύει, γιατί υπάρχει μια σωστή εμπορική ε, ισορροπία μεταξύ όλων των πλευρών που έχουν να κάνουν με τον τομέα. Η ενιαία αγορά είναι μια αγορά που παρέχει, προσφέρει καινούργιες προοπτικές, καινούργιες δυνατότητες, καινούργιες ευκαιρίες τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον δημιουργό ή τον πάροχο υπηρεσιών. Η πολιτική της Ένωσης πρέπει να έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό προς την ανάπτυξη των ε, νόμιμων μέσων προσβάσιμων σε όλους που ευνοούν την καινοτομία, τη δημιουργία. Αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο είναι να εγγυηθούμε μια νομική ασφάλεια στον, ε, στο διαδίκτυο και να αποφύγουμε ε, καταστάσεις άνησης μεταχείρισης μεταξύ της διαδικτυακής και της μη διαδικτυακής υπηρεσίας υπηρεσία. Όπως το υπογράμμισε η Επιτροπή, οι περισσότερες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στοχεύουν βασικά σε ένα εθνικό κοινό ή σε μια ε, ε, πολύ προσδιορισμένη και καθορισμένη γλωσσική ζώνη. Για λόγους για τον οποίο το θέμα δεν είναι να επιβάλλουμε ε, νομικαίους περιορισμούς σε μέσα τα οποία καλύπτουν περισσότερες επικράτειες, περισσότερες γλώσσες, περισσότερες πλατφόρμες, γιατί η ζήτηση είναι πολύ περιορισμένη. Το να επιβάλλουμε μια πανευρωπαϊκή άδεια θα διευκόλυνε την ε, δημιουργία μονοπωλίων από εκείνου που είναι πολύ ισχυροί στην αγορά σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απαρτίζουν πραγματικά τη ραχοκοκαλιά του τομέα των οπτικοακουστικών έργων και των κινηματογραφικών έργων. Πέρα από αυτούς τους άξονες, εργάστηκα γύρω από ορισμένες ιδέες τις οποίες, κατέληξα μετά από ευρύτατες διαβουλεύσεις. Ιδέες πολύ ουσιώδεις για την ε, διαδικτυακή διακίνηση των οπτικοακουστικών μέσων. Πρώτον, διασφάλιση της, της ε, νομικής ασφάλειας για τους συγγραφείς και την ε, πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεύτερον, να επιτευχθεί μια σωστή εμπορική συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων του τομέα με σεβασμό τη χρονολογία των μέσων, τη χρονολογική σειρά των μέσων, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος ταυτοποίησης των οπτικοακουστικών έργων, ε, διεθνές ε, εργαλείο, και για, τις, για τα πολυμέσα και για τα κινηματογραφικά έργα να υπάρχει ένα είδος ε, ταυτοποίησης του DNA των έργων. Θα πρέπει να σεβαστούμε επίσης και το διαδίκτυο, καθοριστικό μέσο για τη διάδοση των έργων και για τον πλουραλισμό των μέσων. Θα πρέπει να σκεφτούμε την προσαρμογή ε, των καθεστώτων που ισχύουν στη χώρα προέλευσης στα νέα μέσα για να αποφύγουμε τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την, ε, την ε, σύναψη συλλογικών συμβάσεων ή αντιπροσωπευτικών συμβάσεων μεταξύ των εκπροσώπων των δημιουργών και των παραγωγών, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει μια αναλογική και εύλογη και δίκαιη αμοιβή για την ε, ε, διαδικτυακή εκμετάλλευση των έργων. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε γρήγορα τη συζήτηση ε, για να δούμε ποιος ΦΠΑ θα επιβάλλεται στις διαδικτυακές και μη υπηρεσίες. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίεργες καταστάσεις που ισχύουν. Θα κλείσω εδώ την συζήτηση και θα ακούσω με μεγάλη προσοχή όλες τις παρατηρήσεις που θα μου επιτρέψουν να ολοκληρώσω και να συμπληρώσω την ε, έκθεση στο πλαίσιο του, χρονοδια... χρονοδιαγράμματος που ανέφερε και ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Καβαντά. Ο λόγος στον κύριο Μπόρις. Ε, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον κύριο Καβαντά για τη θαυμάσια έκθεσή του είναι μια έκθεση η οποία παίζει και συμπληρωματικό ρόλο για να καταδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιγραμμική αγορά πολιτιστικών προϊόντων. Είναι γεγονός ότι οι δημιουργοί στην Ευρώπη έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλες προκλήσεις. Και χάρη στο πολιτιστικό περιεχόμενο αυτός ο χώρος μπορεί να προσεγγίσει όλους τους πολίτες. Ξέρουμε ακόμα ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια στην ενιαία αγορά της Ευρώπης, τεχνολογικά και νομικά εμπόδια, αλλά συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καβαντά. Είμαι εισηγητή γνωμοδότηση στη Νομική Επιτροπή για τα θέματα αυτά και θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με μεγάλο πνεύμα ευθύνη. Θα θέλαμε ότι μια μεριά η πολιτιστική, η καλλιτεχνική δημιουργή να έχουν το δικαίωμα μιας αξιοπρεπούς και λογικής αμοιβή από το σύστημα του διαδικτύου, πρέπει όμως να θυμόμαστε ακόμα ότι και στην Ευρώπη ένα μεγάλο μέρος των ε, κινηματογραφικών έργων εποφελούνται από ειδική χρηματοδότηση. Μέσα στα πλαίσια αυτά γίνονται οι ταινίε μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν επενδύσεις από τους παραγωγούς και αναλαμβάνουν τον κίνδυνο της ενδεχόμενης αποτυχίας ενός ε, φιλμ ή ενός καλλιτεχνικού προϊόντος. Αν όμως γίνει μεγάλη επιτυχία αυτό το φιλμ, θα πρέπει και οι καλλιτεχνικοί δημιουργοί να συμμετέχουν στα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από αυτήν την ταινία όταν διανέμεται στο διαδίκτυο μέσω του διαδικτύου με άλλους τρόπους σε ειδικέ πλατφόρμες του βίντεο επί το βίντεο on demand. Νομίζω θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια υπεύθυνη προσέγγιση και είναι απαραίτητο να ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει ειδικές, ειδικούς κανόνες για την ε, ανταμοιβή των καλλιτεχνικών δημιουργών, λαμβάνοντας πάντα τα ήθη και έθιμα της κάθε ε, χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν λοιπόν πολύ χρήσιμο να υπάρξει μια πρόταση της Κομισιόν για την δίκαια ανταμοιβή των καλλιτεχνικών δημιουργών. Συμφωνώ και με τον κύριο Καβαντά, ο οποίο είπε σήμερα ότι οι άδειε εκμετάλλευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να μην είναι μια αποτελεσματική λύση, γιατί το οπτικοακουστικό έργο αφορά συγκεκριμένα ακροατήρια, εθνικά ή γλωσσικά. Το σύστημα λοιπόν των πανευρωπαϊκών αδειών μπορεί να μείνει μονάχα σε επίπεδο προαιρετικό. Χάρη σε αυτή την έκθεση όμως πιστεύω ότι μπορούμε να επιταχύνουμε το έργο της Επιτροπής ώστε ο δημιουργικός τομέας που λειτουργεί μέσω του διαδικτύου να είναι πιο προσβάσιμος και να μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Αν δούμε λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη, εμείς παράγουμε περίπου 1.200 ταινίε το χρόνο δύο φορές περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά παρόλα αυτά οι πολίτες χρησιμοποιούν κατά 25% τα έργα αυτά. Τα άλλα 75% είναι αμερικάνικα έργα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να αυξήσουμε την προσβασιμότητα των ευρωπαϊκών ταινιών στο διαδίκτυο και θα ήθελα επίσης να πω ότι υποστηρίζω τη δράση του κυρίου Καβαδά και η πρότασή μας είναι να έχουμε και ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την επιγραμμική διανομή των έργων αυτών και πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσει να εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία, πρόκειται για 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλη επιτυχία γιατί θα είναι η Επιτροπή Πολιτισμού που θα προτείνει έτσι νέες λύσεις για το μέλλον που θα κάνουν ακόμα και πιο έντονο το σύστημα αυτό και πιο ισχυρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν και χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα να εκφράσω τη θέση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Βέρετ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τον κύριο Καβαδά για την παρουσίαση της ε, έκθεσής του, του σχεδίου έκθεσής του. μπορούμε να δώσουμε σε ορισμένα σημεία βέβαια ακόμα περισσότερη έμφαση. Είναι σαφές για μένα ότι βρισκόμαστε σε μια κάπως δύσκολη κατάσταση και επομένως θα πρέπει να κάνουμε δηλώσεις σε σχέση με τα δικαιώματα των καλλιτεστικών δημιουργών χωρίς να έχουμε αποφασίσει ακόμα πώς θα θέλουμε να κινηθούμε με το copyright στον ψηφιακό χώρο. Πιστεύω λοιπόν ότι αν δεν έχουμε την απάντηση για όλα αυτά, τουλάχιστον θα πρέπει να μπορούμε να θέτουμε τα σωστά ερωτήματα. Επομένως θα πρέπει να μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα παραδείγματος χάρη μέχρι ποιου βαθμού θα μπορούσαμε να έχουμε μια συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων. Αυτό είναι μια δυνατότητα. Θα πρέπει λοιπόν να εκφράσουμε τη θέση μας με σαφήνεια σε σχέση με τις πανευρωπαϊκές άδειες και τις υποχρεώσεις που συνάπτονται με αυτές τις άδειες. Βέβαια δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε τι θα οδηγήσουν, σε τι θα οδηγήσουν αυτές οι άδειε, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν πολύ πολυδάπανες για μικρά κράτη ή για μικρές γλώσσες. Αν έχουμε, παραγωγικά μία ταινία στα λετονικά, η οποία είναι υποχρεωμένη να έχει μία ε, πανευρωπαϊκή άδεια, τότε για να παιχθεί στην Ισπανία είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουμε τη μετάφρασή της. Αλλιώς δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι λένε στα λετωνικά. Μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε αυτή την μόνο απευθυντική θηρίδα, αλλά αυτό θα εξασφαλιστεί μονάχα αν έχουμε μια σαφήνεια και απλότητα στο νομικό πλαίσιο. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα και για τις ε, ε, οπτικοακουστικές υπηρεσίες όπου έχουμε να κάνουμε με την γραμμική χρήση των προγραμμάτων αυτών και τη μη γραμμική χρήση αυτών των ε, προγραμμάτων, ε, τη μη γραμμική εκπομπή τους. Υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο σύγκληση σε τεχνολογικό επίπεδο μεταξύ εκπομπών και αυτών οι οποίοι βλέπουν αυτά τα προγράμματα μέσα από το ίντερνετ με το σύστημα Video On Demand. Όλα αυτά λοιπόν καλύπτονται από διαφορετικούς κανόνες και διαφορετικές ρυθμίσεις οι οποίες δεν μπορούν να διατηρηθούν με την πολυπλοκότητά του στο μέλλον. Και έχω πολλά προβλήματα στο σημείο 7. Ίσως να είναι πρόβλημα μετάφρασης αλλά στα γερμανικά λέγεται ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα μέτρα ώστε να υπάρχουν και ε, να υπάρχει αποτροπή της δημιουργίας μη εγκεκριμένων πλατφορμών πληρωμής. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει να εμποδίσουμε το παράνομο κατέβασμα από το ίντερνετ. Είναι τόσο μπερδεμένη αυτή η διατύπωση στα γερμανικά, μπορεί να είναι προνομετάφραση, αλλά στα γερμανικά είναι πάρα πολύ ασαφής θα πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε σύμφωνοι σε σχέση με το θέμα της ουδετερότητας του διαδικτύου και της ισότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επομένως, είναι απαραίτητο να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην κινηθούμε σε λαθασμένη κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την ε, ουδετερότητα του διαδικτύου, αλλά επίσης και σε σχέση με το ερώτημα του βαθμού στον οποίο θα, του συστήματος που θα χρησιμοποιήσουμε για να αποφύγουμε τις ε, παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Εγώ βέβαια δεν είμαι υπέρ της ε, ε, παρακολούθησης των επικοινωνιών στο, στο διαδίκτυο. Πρέπει να διατηρήσουμε το δικαίωμα στην ελευθερία της πληροφορίας και της γλώσσης και αυτό είναι απαραίτητο να το διατηρήσουμε από την άποψη της προστασίας, της ελευθερίας, της έκφρασης και της πληροφορίας. Θα πρέπει αντίθετα να προσπαθήσουμε να έχουμε πιο πολλές δυνατότητες νόμιμου κατεβάσματος από το διαδίκτυο με προσβάσιμες τιμές, με προσβάσιμο τίμημα, αυτό θα ήταν μια πολύ σημαντική πλευρά γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν κάποιος βλέπει μια ταινία από τις Ηνωμένε Πολιτείες και το κατεβάζει από το διαδίκτυο, δεν το κάνει για να κάνει κακό στον καλλιτεχνικό δημιουργό, αλλά γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να έχει γρήγορα πρόσβαση σε αυτή την ταινία. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα χρονικά διαστήματα μέχρι ότου είναι διαθέσιμες οι ταινίες στο διαδίκτυο ή με μορφή DVD και κάποιος που θέλει να δει μια ταινία τελικά καταλήγει να χρησιμοποιήσει αυτές τις παράνομες δυνατότητες. Και το ίδιο γίνεται και με την ε, μουσική. Θέλει κανείς να ακούσει ένα μουσικό κομμάτι, δεν έχει καμιά άλλη δυνατότητα να το κάνει με νόμιμο τρόπο και αναγκάζεται πολλές φορές να χρησιμοποιήσει τα παράνομα συστήματα για το κατέβασμα από το ίντερνετ. Και αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αν θέλουμε να εμποδίσουμε την παράνομη χρήση ε, του διαδικτύου για κατέβασμα με το να δημιουργήσουμε περισσότερες δυνατότητε νόμιμου κατεβάσματος από το ίντερνετ και τα μοντέλα τα οποία υπάρχουν, παραγωγή χάρη για τον ε, ήχο καλέσματος στα κινητά τηλέφωνα, μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε ένα πιο εύκολο τρόπο να πληρώνουμε αυτές τις, ε, αυτό το κατέβασμα από το ίντερνετ. Άμα είναι λοιπόν απλά τα, οι διαδικασίες αυτές, είναι ιδιαίτερα εύστοχες και θα περιστήλουν με τον τρόπο αυτό και την, ε, το παράνομο κατέβασμα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά γενικά το δικαίωμα, τα δικαιώματα των καλλιτεχνικών δημιουργών και θα πρέπει να ξέρουμε και ποια είναι η άποψη της Κομισιόν, γιατί πολλές φορές χρειάζεται να περιμένουμε πάρα πολύ μέχρι να φτάσουμε σε μια πρόταση, μέχρι να δούμε την πρόταση της Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Έτσι, αν ξέρουμε κάτι περισσότερο από αυτά που προτίθεται να κάνει η Κομισιόν, μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. Και επίσης πρέπει να θέσουμε και το θέμα της σύγκλησης των τεχνολογιών και υπάρχει το πρόβλημα αυτό το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως ότι οι δημόσιοι ραδιοσταθμοί μπορούν να βγάλουν κάποια κομμάτια στο διαδίκτυο μόνο για μία εβδομάδα και μετά πρέπει να τα αποσύρουν. Αυτό αντιβαίνει και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίντερνετ. Και πολλές φορές είναι υποχρεωμένοι να ζητούν να πληρώνονται πράγματα τα οποία χρηματοδοτούνται ουσιαστικά από το δημόσιο τομέα. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα συζητήσουμε εδώ και ελπίζω ότι μπορούμε να δώσουμε και κάποιες ενδείξεις <clears throat> προς την Κομισιόν για ποια πράγματα θα πρέπει να εξετάσουν περισσότερο στο μέλλον και προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να πάνε για τη μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων και πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Σάρκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Συμφωνώ και εγώ ότι χρειαζόμαστε αυτή την μόνο απευθυντική θηρίδα. Ο κατακαιρματισμός της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων ε, δημιουργεί προβλήματα στους καταναλωτές, στους πολίτες, ε, στην οικονομία μας ε, επιμονή μου βάσεως δεν είναι ακριβώ το ζήτημα που συζητούμε σήμερα, παρόλο που συνδέεται με την επιγραμμική ε, διανομή οπτικοακουστικών ε, έργων. Γι' αυτό και έχει έρθει η ώρα να μπούμε πλέον στον 21ο αιώνα, γιατί τα συστήματα διαχείρισή μα είναι τόσο παροχημένα που ε, θα τα αποκαλούσα μάλλον τροπιαστικά. Τώρα, κάποιες πιο συγκεκριμένε παρατηρήσεις για το σχέδιο. Στην παράγραφο Α, η αναφορά στις τεράστιες προκλήσεις και αυτό ε, έχει σχέση και με άλλε παρατηρήσει που θα κάνω στη συνέχεια. Βεβαίω και υπάρχουν προκλήσει σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των τεχνολογιών. Αλλά α διερωτηθούμε ποιο είναι ο ρόλο των πολιτικών, ε, των νομοθετών και ποιο είναι ο αντίκτυπο τη αγορά. Νομίζω ότι κάποιε βιομηχανίε που αντιμετωπίζουν προκλήσει εντό αγωγικών πρέπει να μάθουν να καιροτομούν. Στην παράγραφο L όπου δεν μπορεί να υπάρχει βιώσιμη δημιουργία ε, και απουσία πνευματικών δικαιωμάτων, προστατεύονται οι δημιουργοί. Και, αυτό, και αυτή είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται και θα βλέπουμε στο, πλαίσιο της ε, απαραίτητης αυτής μεταρρύθμισης ε, που, ε, στην οποία αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι. Είναι σημαντικό να μην κολλήσουμε στο status quo παροχημένων νόμων και να καταλάβουμε ότι με την ε, ανάδυση αυτής της ψηφιακής εποχής κάποιοι φορείς που παλαιότερα ήταν απαραίτητοι για τη διανομή των έργων ενδεχομένως πλέον να μην είναι απαραίτητοι. Ε, αυτός είναι ο αντίκτυπος της ε, ελεύθερης αγοράς και αυτό δεν θα πρέπει να πλήξει ούτε τους παραγωγούς, τους δημιουργούς, ούτε τους καταναλωτές. Είναι μια υγιής μετάβαση στην σύγχρονη κοινωνία. Στην παράγραφο όμικρον, όπου λέμε ότι η αποτελεσματικότητα των ε, φορέων κοινή ε, διαχείρισης πρέπει να βελτιωθεί με τη διαφάνεια κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε και την ε, βελτίωση των υφιστάμενων δομών και όχι μόνο να εξετάζουμε τα παλιότερα συστήματα. Τώρα να υπάρχει και μεταρρύθμιση πέρα από τα παλιότερα συστήματα. Μετά στο Q χρονολογική διάσταση των μέσων επιτρέπει μια ισορροπία και προχρηματοδότηση των έργων. δεν νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτό το, ε, το παράθυρο με κάθε κόστος. Αυτό σου γινόταν παλιότερο, όταν είχαμε τα μονοπόλια που δεν μπορούσε να, να, να υπάρξει παραγωγή ε, και μάλλον πρόσβαση σε τέτοια έργα χωρίς ε, κάποιον μεσάζοντα. Έχει όμως παρέλθει αυτή η εποχή. Τα release windows, αυτό το, το παράθυρο χρήσης, είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο και δεν πρόκειται για πολιτική νομική απόφαση. Μετά στο 3. Και πάλι για αυτές τις στηρίδες αξιοποίησης πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μπλοκάρουμε έτσι την ε, επιγραμμική εκμετάλλευση και να μην καθίσταται πιο ευέλικτη αυτή η αξιοποίηση. Αναφέρεται εδώ ως πολιτική απόφαση, όμως αυτό δεν είναι σωστό. Πρόκειται για επιχειρηματική απόφαση. Δεν πρέπει να συγχαίουμε λοιπόν τον, τον, την πολιτική και ε, την οικονομική ζωή σε αυτό το τομέα. Κάτι άλλο, ένα άλλο ερώτημα που έχω εδώ για το 11 τα καλύτερα μέσα για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς αμοιβή για τους ε, δικαιούχους για, είναι η ενσωμάτωση των ε, παραγωγών και ερμηνευτών. Μια κοινή σύμβαση δηλαδή. Όμως ε, εδώ πρέπει να δούμε τι έχουμε επιτάπητο και θα πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα τι ρόλο θα έχει να δραματίσει ο πολιτικός τύπος και τι ο επιχειρηματικός. Ας είμαστε λοιπόν ως τον πιο φιλόδοξοι ούτως ώστε να δίνουμε πρόσβαση και στους Ευρωπαίους πολίτες και όμως σε πολίτες άλλων χωρών για να γίνουν τα οπτικοκοστικά έργα πιο προσβάσιμα, πιο οικονομικά και να ξέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και άλλοι πολίτες τι έχουμε να προσφέρουμε στο πολιτιστικό επίπεδο για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Το έργο μα λοιπόν θα πρέπει να αντακατοπτρίζει αυτά τα σημεία στο σχέδιο. Ευχαριστώ. Αντιπρόεδρος Μπίσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 28% μερίδιο στον παλιό αναλογικό κόσμο. Μόνο 2% στον ψηφιακό κόσμο που είναι η νέα τεχνολογία. Ξέρετε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει μέσα σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αν δείτε την οπτικοακουστική αγορά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σαφές ότι οι πιο, παρα... οι δημιουργικές εταιρείες και οι μικρές εταιρείες εξαρτώνται από τους τωρινούς ε, σταθμούς και παραγωγούς πολιτιστικών ε, προϊόντων και υπόκεινται στις επιταγές αυτών των παραγωγών. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήττει. Ξέρουμε ότι είναι πολλές φορές ε, υποχρεωμένοι να παρέχουν τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο η καλλιτεχνική δημιουργή χωρίς πρόσθετη ανταμοιβή. Για, την, ε, για το ραδιοφωνο, την τηλεόραση και το κινηματογράφο σιγά σιγά συνενώνονται οι μορφές παραγωγής και παροχής προς το κοινό ώστε να είναι όλο και πιο δύσκολο για τους ανεξάρτητους παραγωγούς να μπορέσουν να επιβιώσουν. Η κατάσταση λοιπόν και των καλλιτεχνικών δημιουργών και των μικρών εταιριών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εξάρτησή τους από τα μεγάλα συγκροτήματα ώστε να μπορέσει να εξασφαλιστεί ότι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα στο διαδίκτυο. Και αυτό φυσικά σημαίνει και την ε, καλύτερη πρόσβαση των χρηστών. Ο χρήστης είναι όχι μονάχα καταναλωτής αλλά και παραγωγός γιατί η ίδια η ψηφιακή επανάσταση οδηγεί σε μια επανάσταση σε σχέση με τα συστήματα ανταμοιβή των καλλιτεχνικών δημιουργών. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε λοιπόν μέσα στα πλαίσια και της προστασίας των δεδομένων και της ουδετερότητος του δικτύου. Θα ήθελα τώρα να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με το σχέδιο γνωμοδότηση του κυρίου Καβαντά για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Καβαντά. Εσείς έχετε πράγματι κάνει μια πολύ καλή έκθεση και είναι μια πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση. Αναφέρεται ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Εγώ αυτό το οποίο κατανοώ είναι ότι με την εξέλιξη των δικαιωμάτων των πνευματικών θα πρέπει να να την προσαρμόσουμε και αυτή στον ψηφιακό κόσμο. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε όσα έχει η ρύθμιση για τον αναλογικό κόσμο. Θα σας δώσω το παράδειγμα ενός φίλου μου, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει όταν αλλάζει όταν, αλλάξαμε από τις άμαξες στα αυτοκίνητα, δημιουργήθηκαν και νέοι κανόνες κυκλοφορίας και δεν μείναμε μονάχα στους κανόνες κυκλοφορίας των αμαξών. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει νέο σύστημα για την ε, ε, ταυτοποίηση και την ταξινόμηση των έργων. Παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, αν πει κάποιος ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα, στις επιστολές που έχουν γραφεί στο παρελθόν, αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα νομικά. Κύριε Καβαντά, επίσης, εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ε, μπλοκαρίσμα, δεν μπορεί να υπάρξει ε, λύση μόνο με τον μπλοκάρισμα ορισμένων ιστοσελίδων στο ίντερνετ, η οποία απορρίπτεται από τους περισσότερους στη Γερμανία. Νομίζω ότι επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε με ποιο τρόπο, με τρόπο θα μπορούμε να έχουμε εταιρείε οι οποίες απλώς κάνουνε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή ή για υπολογισμό τελών και δεν οδηγούν σε παραγωγή ή παροχή νέων ε, στοιχείων πολιτιστικών. Πρέπει να μπορέσουμε επίσης να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει και μια ενεργή συμμετοχή των νέων στις δραστηριότητες αυτές, γιατί είναι ως παραγωγή και ως καταναλωτές αυτοί οι οποίοι κυριαρχούν στο ίντερνετ. Αυτό ήταν πολύ θετικό. Ευχαριστώ κύριε Μπίσκι. Και τώρα η κυρία Μακλάρκεν. Ευχαριστώ. Μιας και ήδη έχουμε συζητήσει τη συμβολή των καινοτόμων πολιτιστικών επιχειρήσεων, πιστεύω ότι ο τομέας αυτός είναι κρίτιμος για την, κρίσιμος για τη διατήρηση της ε, ποικιλία και της πολυμορφίας και χρειάζεται πραγματικά μια πλατφόρμα για, την, ε, για τις ταινίες και άλλα μέσα και να ε, υπάρχει επίσης αυτή η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στα πολιτιστικά, πολιτισμικά, στα έργα του πολιτισμού. Ε, νομίζω πολλές καλές υποδείξεις έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο για το πώς θα ανταποκριθούμε στις διάφορες προκλήσεις. Ε, φυσικά υποστηρίζω το σύστημα πληρωμής όπως αυτό που ισχύει για τα μηνύματα ε, επίσης ε, μια μικροχρέωση για τις υπηρεσίες streaming. Επίσης να υπάρχει ένας μηχανισμός εμπλοκής εκείνων των ιστοσελίδων οι οποίες παραβιάζουν τον νόμο. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν νόμιμα μέσα στη διάθεσή μας για, να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα. Κύριε Καβαδό Αναγνωρίζει βέβαια ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν νομικά προσκόμματα στη διαπραγμάτευση ε, συμφωνιών ε, που θα ισχύσουν σε πολλαπλές επικράτειες ή που θα έχουν εφαρμογή σε πολλαπλά πολυμέσα. Θα πρέπει επίσης να, υπάρχει, να εξασφαλιστεί η ελευθερία των συμβάσεων, να υπάρχει κάποια εξασφάλιση της διανομής των έργων τους και θα πρέπει να προσδιορίσουμε σαφώς ε, ποια δικαιώματα θα, για ποια δικαιώματα θα απαιτείται άδεια χρήσης. Το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται στον σκοπό του. Ε, θα πρέπει το copyright να μην γίνεται τόσο ακριβό ώστε να μην εκπληρώνεται ο σκοπός του στο τέλος. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διάφοροι θεσμοί πολιτιστημικής κληρονομιάς θα μπορούν πραγματικά να διαθέτουν ε, τα έργα που έχουν στη διάθεσή τους, όπως για παράδειγμα η ε, Βρετανική Ταινιοθήκη και παρόμοιοι οργανισμοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Φερχάιεν. Äh, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καβαντά ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχει αντιμετωπίσει και νομίζω ότι η εκθεσή του είναι πολύ καλή και πολύ καλά διορθωμένη. Και πράγματι είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι πάρα πολλά και ε, καλύπτουν ένα πάρα πολύ ευρύ τομέα. Είναι απαραίτητο η Κομισιό να μας δώσει περισσότερο υλικό και κυρίως να συνδέσει καλύτερα όλα αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει κάπως να αντιμετωπιστούν από κοινού. Συζητήσαμε πρόσφατα για το θέμα των Open Works και η Κομισιόν έχει κάνει κάποιες προτάσεις για τα θέματα αυτά. Έχουμε συζητήσει για το copyright. Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο από θέματα τα οποία συνδέονται πάρα πολύ άρρηκτα μεταξύ τους και δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το ένα χωρίς να λάβουμε υπόψη και τις ε, επιπτώσεις που θα προκύψουν για τα άλλα. Το Open Works είναι μια νέα πρωτοβουλία για το copyright, αλλά φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μαζί με το copyright. Όλα αυτά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μονάχα σαν μια δέσμη μέτρων και μας έρχονται από την Κομισιόν ένα-ένα στην περίπτωση της έκθεσης του κυρίου Καβαντά υπάρχει το, η προσπάθεια του εισηγητή να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα αλλά σίγουρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη στενή σύνδεση όλων των θεμάτων αυτών για τις ε, εταιρείες χάρη που κάνουν συμπιλήσεις. Εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο γιατί έχουμε πάρα πολλές υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να γίνει πιο εύκολο να μπορέσει κανείς να αποκτήσει τα δικαιώματα για τη συμπίληση έργων και να κάνει αποτρεπτική την ε, παράνομη χρήση αυτών των ε, έργων. Το σημείο 7 αναφέρει ότι δεν πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε πλατφόρμες πληρωμής εάν δεν είναι νόμιμα αυτά τα έργα τα οποία χρησιμοποιούνται, η χρήση αυτών των έργων, εγώ νομίζω ότι πρέπει να το γυρίσουμε ανάποδα, ότι αυτές οι πλατφόρμες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει καταχρηστική ε, πρόσβαση σε, σε κάποια έργα. Όχι λοιπόν να μην όχι να εμποδίζουν για όλους την πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες, αλλά οι πλατφόρμες αυτές να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει πρόσβαση εάν δεν είναι νόμιμη η πρόσβαση στα έργα αυτά. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνουμε για τα για άλλες πλατφόρμες. Όταν είναι κάτι, όταν είναι σαφές ότι μια πλατφόρμα παραβιάζει το δίκαιο, τότε αυτή η πλατφόρμα θα πρέπει να αφαιρεθεί από το δίκαιο, από το διαδίκτυο, όπως γίνεται για ιστοσελίδες ε, παιδικής πορνογραφίας. Δεν μπορεί λοιπόν να επιτρέψει κανείς την ύπαρξη τέτοιων πλατφορμών. Κάποιος ο οποίος πουλάει κάτι το οποίο δεν του ανήκει είναι παράνομος, αν αυτό είναι ένα πολιτιστικό προϊόν, ένα ε, έργο ή ένα μουσικό κομμάτι. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να επιβάλλουμε περιορισμούς ή να απαγορεύσουμε τελείως αυτά, τα, αυτές τις πλατφόρμες. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι το θέμα της ε, καλύτερης ε, μορφής συντονισμού. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα, όπως ελέγχθη, να υπάρχουν πιο πολλές νομικές νόμιμες δυνατότητες ώστε να μπορεί κανείς με πιο ευτελές τίμημα να μπορέσει να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε όλα αυτά ώστε να έχουμε και μια καλύτερη πρόσβαση στα προϊόντα αυτά. Δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια κοινωνία του copy and, copy and paste, ώστε όλοι να αντιγράφουν από όλους χωρίς να παίρνει ποτέ ο δημιουργός ένα team αυτό. Ούτε θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα με κίνον όπως το παρελθόν όπου χωρίς ένα ισχυρό με κίνα δεν μπορεί κανείς να παραγάγει ένα πολιτιστικό αγαθό πρέπει να καταλήξουμε σε ένα βιώσιμο σύστημα όπου αυτοί οι οποίοι παράγουν το πολιτιστικό περιεχόμενο να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε ένα ισχυρό σύστημα copyright το οποίο όμως να είναι προσαρμοσμένο στο διαδίκτυο και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν και κατακαιρματισμοί σε επίπεδο εθνικού περιεχομένου ή γλωσσικού περιεχομένου Θέλουμε ένα σύστημα το οποίο θα εξασφαλίσει ότι υπάρχει η ροή των κονδυλίων, των ε, τελών και των αμοιβών σε αυτούς οι οποίοι είναι οι καλλιτεχνικοί δημιουργοί και να επιτρέψει επίσης και στους ερμηνευτές όπως είναι οι ηθοποιοί να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν. Ξέρουμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε πάντα ενδιάμεσους, ενδιάμεσες εταιρείες κτλ. Αλλά θα πρέπει όλους αυτούς οι οποίοι προβαίνουν στην ανα, ε, παρουσίαση έργων ή στη συμπίληση έργων να τους περιορίσουμε σε σχέση με τη δυνατότητα που μπορούν να έχουν να παίρνουν τη μερίδα του λέοντος από όλα, από τα αγαθά αυτά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα συντονισμό, δεν αυτό απαιτεί μια κεντρική υπηρεσία, αλλά να έχουμε μια κεντρική ε, πύλη πρόσβασης για το νόμιμο κατέβασμα, κατεβάσματος των έργων. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και συγχαρητήρια στον κύριο Καβαντά για την εξαιρετική του έκθεση. Πολλά υπόθηκαν ήδη και σε πολλά συμφωνώ. Δύο-τρεις παρατηρήσεις έχω μόνο για την μονοπευθυντική θηρίδα, το One Stop Shop και για την εύκολη πρόσβαση. Γιατί είμαι πεπισμένος ότι αυτό είναι το κρίσιμο σημείο και η κύρια πρόκληση είναι η εύκολη πρόσβαση για τους καταναλωτές σε νομικό υλικό υψηλής ποιότητας. Αν θέλει κάποιος, σε παράδειγμα, να ε, δει μια ταινία στο διαδίκτυο, είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό μέσω ε, ενός, μιας, ενός παράνομου στο τόπο παρά να βρει έναν νόμιμο πάροχο. Αυτή είναι η αλήθεια. Επομένως, μόνο με το να έχουμε μια εύκολα προσβάσιμη, νόμιμη συγγνώμη, ε, λύση θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση. Και πέρυσι είχαμε την, ε, αυτή η γεωμετρική αύξηση των παράνομων ε, θεάσεων, αν θέλετε, μειώθηκε πάρα πολύ γιατί υπήρχαν και πολλές οργανώσεις που παρατηρούσαν τι συνέβαινε στο διαδίκτυο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή ο ίδιος ο τομέας να μπορέσει να παρέμβει και εμείς να τους βοηθήσουμε για να αναπτύξει αυτό το περιεχόμενο το νόμιμο και υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, είμαι σίγουρος ότι αυτή η νόμιμη πλατφόρμα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και για πολίτες εκτός της εθνικής επικράτειας, γιατί μιλάμε και διαφορετικές παραδόσεις ή έθιμα, αλλά πρέπει να έχουμε ως προτεραιότητα την ύπαρξη μιας πραγματικής ε, ενιαίας αγοράς, ενιαίας ε, ψηφιακής αγοράς. Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν λύσεις σε αυτό το τομέα. Πρέπει, Θέλω να βρούμε ε, εναρμονισμένα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Αρκετοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο One Stop Shop ή τουλάχιστον στη μείωση των διαδικασιών, στον περιορισμό των διαδικασιών για την ε, κατοχήρωση δικαιωμάτων. Αυτό είναι μια δεύτερη προτεραιότητα. Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε εκ νέου τον ε, τροχό, αλλά ε, συστήματα που ήδη λειτουργούν καλά και υφίστανται ήδη, για παράδειγμα, στις σκανδιναμικές χώρες, μπορούν να αξιοποιηθούν. Πολλοί συνάδελφοι συμφωνούν από αυτού. Πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε πιέσεις. Και τέλος, συνάδελφα Καβαδά, πολύ καλά τα είπε στο σημείο 14, ομοιωμένος ε, συντελεστής ΦΠΑ, ε, για να μην υπάρχουν να καταργηθεί αυτή η ανισορροπία μεταξύ ψηφιακού και μη ψηφιακού υλικού. Συμφωνώ πολύ από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ας δούμε αν έχουμε εκπροσώπους από την Επιτροπή, από την ε, Εσωτερική Αγορά. Ε, η κυρία Βόλβη είναι εδώ. Νομίζω δεν είναι εδώ. Αν όχι από την Διεύθυνση Παιδεία και Πολιτισμός, ο κύριος Τζόι. Α, απεργεί η Επιτροπή σήμερα. ζωή, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, δικό μου σφάλμα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που μπορώ να πω εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης ε, Πολιτισμός και Εκπαίδευση πάνω σε αυτήν την ισορροπημένη έκθεση η οποία λαμβάνει υπόψη της, ε, ε, της, τις διαφορετικές εκφάνσεις της διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα το ζήτημα της πειρατείας το ζήτημα της προστασίας ε, των δικαιούχων, καθώς επίσης και το ζήτημα της προστασίας της πολιτισμικής ε, πολυμορφίας. Πάνω σε αυτό, πιστεύω πως είναι χρήσιμο όχι μόνο να επιμείνουμε ε, στο ζήτημα της κληρονομιάς, της κινηματογραφικής κληρονομιάς, αλλά και στην πραγματική προσφορά που υπάρχει σήμερα και η οποία πρέπει να ιδωθεί. Θα πρέπει να αναπτύξουμε νόμιμους τρόπους διάθεσης των έργων προς τους ε, πολίτες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ε, νόμιμης διάθεσης ε, και την ανάπτυξη υψηλού ανταγωνισμού. Το είδαμε αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος ε, Media για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα. Είναι αρκετά δύσκολο να να ενταχθεί κανείς στις διάφορες ευρωπαϊκές πλατφόρμες. Είναι δύσκολο να θεσπιστεί, να κατοχυρωθεί ε, ένα σήμα, αν θέλετε, έναντι των διεθνών μεγάλων πλατφορμών, το iTube και πολλές άλλες που όλοι γνωρίζετε. Ε, θα πρέπει εμείς από την πλευρά μας να ευνοήσουμε ένα ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο διευκολύνει αλλά και να δώσουμε και ενισχύσεις γιατί πραγματικά απαιτούνται κρατικές ενισχύσεις που να διευκολύνουν την ανάπτυξη τέτοιων ευρωπαϊκών πλατφορμών οι οποίες να διαθέτουν και τα ευρωπαϊκά έργα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Εξίσου σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής της ε, οδηγίας ε, για τα οπτικοακουστικά έργα και τις υπηρεσίες. Ο συνάδελφος εδώ από την Γενική Διεύθυνση της Κοινωνίας Πληροφοριών που ασχολείται με αυτή την προβληματική θα επιμείνει και εκείνος στο γεγονός ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν πραγματικά και αποτελεσματικά μέτρα έτσι ώστε οι διάφορες πλατφόρμες των βίντεο on request να, να λειτουργήσει σωστά για να μπορέσει να διατεθεί το ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Ε, υπάρχουν ένα σωρό έργα τα οποία δεν διατίθενται. Ε, εν πάση περιπτώσει, ήδη έχει υπάρξει ένα δημόσιο εργαστήριο πάνω στο θέμα, μια μελέτη attentional είναι η επωνυμία του, της, ε, του consortium, της κοινοπραξίας που διεξήγαγε αυτή τη μελέτη για αποτελεσματικούς τρόπους διάθεσης και προώθησης ε, των ευρωπαϊκών έργων μέσω μιας πλατφόρμας. Θα είναι χρήσιμο ασφαλώ να υλοποιηθεί αυτό, γιατί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε μια προπαρασκευαστική ενέργεια για την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών έργων, που στόχο έχει να δοκιμάσει, να τεστάρει νέες μορφές ε, διάθεσης ε, των έργων, ε, διάθεσης που θα μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα σε πολλές εθνικές επικράτειες. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια χρονολογική σειρά. Τα έργα βγαίνουν πρώτα σε μία επικράτεια και μετά διαδοχικά περνούν ε, σε άλλες. Ε, ε, το Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει λοιπόν αυτόν τον τρόπο σύγχρονης διάθεσης σε πολλές επικράτειες και σε διαφορετικές πλατφόρμες. Έχουμε διαθέσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται να προκηρυχθεί και ε, μια πρόσκληση ενδιαφέροντος τον ε, Απρίλιο για να φέρουμε και μια διαφάνεια στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι πραγματικά πρόκειται για εξαιρετικό έγγραφο. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Αλλά ίσως ο συνάδελφος ο Αγάλτ έχει να πει κάτι παραπάνω. Παρακαλώ μόνο μία παράκληση. Για να είμαστε συγκεκριμένοι και ειδικοί, θέλω να σας ρωτήσω εάν πραγματικά εκφράζετε τη γνώμη της Επιτροπής. Για να είμαστε συγκεκριμένοι. Απάντηση. Πιστεύω ότι πράγματι πρόκειται για μια ισορροπημένη θέση. Βεβαίως υπάρχουν αποχρώσεις, ε, ε, τα γνωρίζετε πώς λειτουργούν τα πράγματα συνήθως, αλλά απευθύνομαι και στους συναδέλφους εδώ από την ε, Γενική Διεύθυνση της Κοινωνίας των Πληροφοριών, αν θέλουν να πούν κάτι άλλο, αν πιστεύουν ότι αξίζει κάτι να προσθέσουν, να σχολιάσουν. Πέρα από την δύσκολη θέση, γιατί ήταν η Γενική Διεύθυνση Αγοράς η οποία τέλος πάντων προείστα, προείστατο και εκείνη θα έπρεπε να λάβει το λόγο. Του του τουλεχθέντος όμως. Ε, εντάξει, δεν κατάλαβα καλά τι εννοείτε. Τέλος πάντων, σα ευχαριστώ ε, για, για αυτά που είπατε. Εμεί θέλουμε πραγματικά να ξέρουμε ποια, επακριβώς ποια είναι η θέση της Επιτροπής, γιατί έτσι διευκολύνεται το έργο ολόκληρη της Επιτροπής μας και συγκεκριμένα του συναδέλφου του κυρίου Καβαντά, στον οποίο και μάλιστα δίνω ευθύ αμέσω το λόγο για τα, για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, αυτό το οποίο με ενθαρρύνεται να κάνω είναι να συνεχίσω μια εργασία ε, ένα έργο στο οποίο δεν υπάρχει αντίστοιξη, όπως θα λέγαμε, με μουσικούς όρους. Γενικά πιστεύω ότι το θέμα αυτό είναι ένα σύστημα, ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με μεγάλη ταχύτητα. Βέβαια ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και έντονη συζήτηση. Έχω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν συμβάλει στα θέματα αυτά, με τις απόψεις τους ή με τις πληροφορίες τους, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και καταδεικνύουν ένα τουλάχιστον πράγμα, ότι αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι να καταλήξουμε σε μια κάπως πρωτότυπη θέση. Από τη μία πλευρά, από τη μία πλευρά θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στο έργο μας, να μην καταλήγουμε σε κείμενα τα οποία πάνε κατευθείαν στην στον κάλαθο των αχρήστων. Επομένως θα πρέπει να μας εμπνέει ο ρεαλισμός. Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τους άλλους εμπλεκομένους. Δεν πρόκειται για ένα νομοθέτημα το οποίο θα παραγάγει περιεχόμενο καλλιτεχνικό ή συστήματα διανομής. Πρέπει όμως συγχρόνως να έχουμε και μια πολιτική σκέψη με την ευγενή έννοια της πολιτικής σκέψης για να θέσουμε ένα σωστό πλαίσιο υπέρ και των καλλιτεχνικών δημιουργών και υπέρ και των χρηστών ή καταναλωτών. Ένα πολύ απλό θέμα θέλω να, ένα πολύ απλό σημείο θέλω να υπενθυμίσω ότι η πρόσβαση, η ελευθερία πρόσβασης στα νέα μέσα, τα ηλεκτρονικά, δεν έχει να κάνει με την καλλιτεχνική παραγωγή, αλλά με τη διανομή των καλλιτεχνικών αγαθών. Και δεν υπάρχει καμία ζωντανή κουλτούρα, ζωντανό πολιτιστικό τομέα, χωρί <clears throat> τα λαμβάνει κανεί υπόψη τα οικονομικά στοιχεία. Ή έχουμε το αμερικανικό σύστημα το οποίο ελέγχει όλα τα ε, στοιχεία της καλλιτεχνικής παραγωγής και η πιο προχωρημένη κατά κάποιο τρόπο πιο ψαγμένη καλλιτεχνική δημιουργή της Αμερικής ζητούν να υπάρχει ένα πιο διαφοροποιημένο σύστημα όπως το ευρωπαϊκό που επιτρέπει σε όλους να έχουν μια παρουσία. Πιστεύω λοιπόν ότι εμείς θα πρέπει να διατηρήσουμε τη μεγάλη πολιτιστική μας πολυμορφία, αλλά θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο επιτρέπει στην διατήρηση αυτής της πολυμορφίας να έχουμε ένα πλαίσιο και συγχρόνως να μην συγχαίουμε το σύστημα αυτό οικονομικής οργάνωσης του πολιτιστικού τομέα με το σύστημα διανομής το οποίο είναι αυτό το οποίο εξασφαλίζει την πρόσβαση σε όλους. Δεν θέλουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέψει την εισβολή των αμερικανικών προϊόντων σήμερα και αύριο από την Ασία κτλ. Πρέπει να προστατεύσουμε λοιπόν την πολιτιστική μας ε, πολυμορφία και να την διατηρήσουμε. Επίσης, Νομίζω ότι κάποιος, η κυρία Κάμεφερτ έκανε μία παρατήρηση που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, ότι θα πρέπει να ξαναεξετάσουμε κάποτε αυτά τα οποία έχουν θεσπιστεί νομοθετικά στο ευρωπαϊκό σύστημα για τα μέσα ενημέρωσης. Μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή όπου τα νέα οπτικοακουστικά έργα έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά συστήματα διανομής. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένας εξυγχρονισμός αυτού του κειμένου των νομοθετικών ευρω... κειμένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως και μια απλοποίηση. Και ένα τελευταίο στοιχείο, τώρα μπαίνω στις λεπτομέρειες των απαντήσεων, αλλά φυσικά οι, με τους κοιόδης εισηγητές θα επανέλθω σε μια πιο ευρεία διαβούλευση. Εγώ προσωπικά είμαι διστακτικός για όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με απλοποίηση. Θα ήθελα τουλάχιστον να τα δω με κάποια επιφύλαξη. Στη χώρα μου, κάποια στιγμή στη ζωή μου, ήμουνα υπεύθυνο μιας μεγάλης εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών. Δεν μπορεί κανείς και να παράγει έργα και να ψάχνει να βρει ερμηνευτές και να κάνει και την ε, οικονομική διαχείριση. Πρέπει να δούμε λοιπόν όλους αυτούς ως σύνολο. Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό το οποίο λέμε παράθυρα. Όχι για να εμποδίσουμε την πρόσβαση, αλλά για να δημιουργήσουμε νέους οικονομικούς πόλους οι οποίοι δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Αν βάλετε ένα έργο στην αγορά του σινεμά και συγχρόνως στην τηλεόραση, τότε δεν θα έχετε χρηματοδότηση. Γιατί ποιο χρηματοδοτεί αυτή τη στιγμή το σινεμά. Κυρίω η τηλεόραση. Το ίντερνετ δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ακόμα το σινεμά. Δεν πρέπει λοιπόν να καταστρέψουμε συστήματα τα οποία λειτουργούν για να βρούμε νέες λύσεις. Διαπιστώνω πάντως και πάλι ότι όλοι μας ενδιαφερόμαστε, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικές φόρμουλες για να το επιτύχουμε, να προστατεύσουμε τον ακουστικό τομέα είναι κάτι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη και εκμεταλλεύουμε αυτή την ευκαιρία ότι θα πρέπει να βρούμε στην έκθεση αυτή τον τρόπο να τονίσουμε το πώς τα πολιτιστικά θέματα δεν μπορεί να θεωρούνται ως μονάχα μια δευτερεύουσα απόφυση για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρόσχημα της επικουρικότητας. Θα πρέπει να βρούμε πιο ισχυρά συστήματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα γιατί σε μια χρονική στιγμή που η κοινή γνώμη ουσιαστικά απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη βλέπει σαν οπισθοδρομική, ο κυριότερος τρόπος να πλησιάσουμε τους ανθρώπους είναι τα οπτικοακουστικά έργα. Θέλω λοιπόν να σας ε, να συμμεριστώ αυτή την άποψη μαζί σας ότι είναι κατεπήγον να υπάρξει μια μεγαλύτερη συνοχή στην Ευρώπη τονίζοντας όλα αυτά τα οποία μας ενώνουν και αυτό θα γίνει με την υποστήριξη της ε, οπτικοακουστικής δραστηριότητας. Έχουμε χώρες στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν κινήματα αντίδρασης. Επομένως δεν πρέπει να δούμε τα πολιτιστικά θέματα σαν ένα διακοσμητικό κομμάτι της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Ξέρω ότι υπάρχει αρχή της επικορικότητας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε μόνη την επικορικότητα να αλωνίζει. Είναι τέτοιε οι στιγμές που πρέπει να έχουμε μια στεναρή στάση για τα οπτικοακουστικά σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Καβατά. Υπενθυμίζω ότι σχετικά με αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 12 Απριλίου στις 12 και θα ψηφίσουμε στις 19 Ιουνίου. Σημείο 9. Τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης του πρωινού. Χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινοί κανόνες για την ελευθερία κυκλοφορίας θα σημάστε τη μακρά ιστορία αυτού του φακέλου. Η Επιτροπή Λίμπε ζήτησε την άδεια να επεξεργαστεί μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για την ελευθερία των μέσων και την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Η Επιτροπή Πολιτισμού το αμφισβήτησε γιατί θεώρησε τον εαυτό υπεύθυνο, τον εαυτό της υπεύθυνο για το για τον τομέα αυτό, για το θέμα αυτό. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θεώρησε ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο θέμα θεμελιωδών ελευθεριών για τα μέσα πληροφορίες. Η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε εν τέλει να δώσει στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να προχωρήσει. Ο εισηγητής είναι ο κ. Βέμπερ. Η δική μας Επιτροπή θα υποβάλει γνωμοδότηση. Νιγκάρσκι είναι η συγητή μα. Θα μας παρουσιάσει το σχέδιο σήμερα, θα ψηφίσουμε το Μάιο. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 12 Απριλίου, ώρα 12. Μιγκάσκι. Κύριε Μιγκάρσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα είμαι πολύ σύντομος λοιπόν και προσπαθήσω να συνοψίσω. Το έγγραφό μου παρτίζεται από τέσσερα άθρα. Στο πρώτο, στους την προσοχή στην βελτίωση ε, του ρόλου ε, των ελεύθερων και ανοιχτών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει λοιπόν αυτό να το ε, τονίζουμε, ότι πρέπει να είναι και ελεύθερα και ανεξάρτητα τα ΜΜΕ. Δεύτερον, Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ε, τον απογραμμίζουμε τον ρόλο των δημοσίων μέσα μαζική ενημέρωση. Βεβαίω με κάθε σεβασμό προ τα ε, ιδιωτικά μέσα μαζική ενημέρωση, μου φαίνεται ότι τα δημόσια μέσα έχουν και αυτά ένα σημαντικό ρόλο να διδραματίσουν. Και εμεί ω Επιτροπή Πολιτισμού θα πρέπει να τονίζει ε, τον ρόλο αυτών των μέσων. Βεβαίως και συνεργασία πάντα και με τα ιδιωτικά. Τα σημεία 3 και 4 αφορούν τα όσα μόλις συζητήσαμε. για την έκθεση του κυρίου Καβαντά. Δηλαδή υπογραμμίζουμε την ελευθερία του διαδικτύου και των διαδικτυακών μέσων καθώς και των επιγραμμικών πληροφοριών, η πληροφόρησης μάλλον. Αυτά εν συντομία τα κύρια σημεία που συμπεριέλαβα στην έκθεσή μου. Σας ευχαριστώ πολύ και βεβαίως είμαι στη θέσή σας. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Μέντες Τεβάλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπενθυμίσω τη σημασία και το ευαίσθητο του θέματος αυτού που μας απασχολεί. Οι κοινωνίες είναι πιο ελεύθερες βέβαια ότι είναι υγιή τα μέσα ενημέρωσης και όταν αντανακλούν την πολυμορφή απόψεων στις ε, κοινωνίες αυτές. Δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο μας έχει, δώσει, εκδώσει μια σειρά αποψηφίσματα για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σχέδιο γνωμοδότηση τώρα του κυρίου Μικάλσκι, εγώ θέλω καταρχήν να συμφωνήσω στις γενικές γραμμές του, διότι πράγματι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους τους δημοκράτες. Θέλω κατά τα άλλα να πω ότι ίσως αυτή η γνωμοδότηση θα μπορούσε να είναι λίγο πιο φιλόδοξη σε σχέση με το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να φροντίσει και να εξασφαλίσει για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι η συζήτηση για ένα πιο έντονο ρόλο της Κομισιόν είναι απόλυτα απαραίτητη. Γιατί όταν μπαίνει μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προηγουμένως έχει περάσει από αυστηρές προδιαγραφές, δεν υπάρχει τόση επαγρύπνηση αφού γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω επίσης να ζητήσω από την Κομισιόν να υποστηρίξει την πολυμορφία των μέσων ενημέρωση σε χώρε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου λόγω δικτατοριών είναι δύσκολο ή σχεδόν αδύνατο να υπάρχει αυτή η πολυμορφία. Υπάρχει και ένα θέμα τύπου, ίσως θα ήταν καλύτερα να εγγράψουμε αυτό το σημείο σε μια μεταγενέστερη παράγραφο, γιατί η έκθεση την οποία συζητούμε αφορά τα πρότυπα της ελευθερίας του τύπου και των μέσων ενημέρωσης μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο λόγος την κυρία Κάμερβερτ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ μπορώ να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο συναδελφός μου και εγώ πιστεύω ότι το πρώτο σημείο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην γνωμοδότηση βεβαίως είναι σωστό να αναφερθεί αλλά δεν πρέπει να βρίσκεται στο σημείο αυτό αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι πώς θα εξασφαλίσουμε ότι ισχύουν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Επομένως το άρθρο αυτό βρίσκεται ίσως σε λαθασμένη θέση στην έκθεση ακόμα και αν είναι ορθό το περιεχόμενό του. Πάντα έχουμε πολύ καλές σχέσεις μέσα στην Επιτροπή μας, αλλά εδώ πρέπει να πω στον κύριο Μιγκάλσκι ότι είμαι απογοητευμένη με αυτά τα οποία περιέχει η γνωμοδότηση Έχουμε κάνει τουλάχιστον δύο εκθέσεις όπου αναφερόμαστε στα θέματα του πλουραλισμού των μέσων <clears throat> ενημέρωσης. Επρόκειτο για την έκθεση του κύριου Ιβο Μπέλετ σε σχέση με το δημόσιο ραδιόφωνο και το ιδιωτικό ραδιόφωνο και επίσης η έκθεση Lockegaard για, τον, ε, για τη δημοσιογραφία και την ελευθερία άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των καναλιών και των ραδιοφώνων, την ελευθερία των ε, μέσων του έντυπου τύπου, το να μπορέσουμε να αποφύγουμε την υπερσυγκέντρωση σε λίγα χέρια των εφημερίδων. Πώς θα αποφύγουμε λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται σε ορισμένε χώρες που περιορίζεται η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και πώς θα εξασφαλίσουμε την ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων μέσα στα κράτη-μέλη και τα έντυπα και τα κανάλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιλάβαμε στην έκθεση του κυρίου Ιβο Μπέλετ το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ που θα πρέπει να εφαρμόζονται όλα αυτά πρώτα απ' όλα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μονάχα στις υποψήφιες χώρες. Και δεν περιλαμβάνει μονάχα την οργάνωση των καναλιών και των ραδιοφωνικών σταθμών, αλλά και το θέμα της χρηματοδότησής τους. Ξέρω ότι το θέμα της επικουρικότητας παίζει ένα αποφασιστικό ρόλο στα θέματα αυτά, αλλά αν μας ενδιαφέρει να καταλήξουμε σε πρότυπα για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν πολύ πιο απτό και συγκεκριμένο χαρακτήρα από ότι αυτά που βλέπω εδώ στη γνωμοδότηση και θα πρέπει να σταθούμε και στο θέμα της συγκέντρωσης ε, των μέσων ενημέρωσης, της ε, ε, εξασφάλισης της ποιότητος και της αυτονομίας και ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία η γνωμοδότηση αυτή προς την νομική επιτροπή είναι απαραίτητο να υπάρχουν χωρίς να ρίψουμε εκτός το βρέφος με τα ύδατα του μπάνιου του. Να μην καταλήξουμε λοιπόν στο να έχουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή αρχή η οποία υποτίθεται θα τα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Πρέπει όμως να απευθυνθούμε σε αυτό το σύνολο προβληματικής. λόγος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως είπε η κυρία Καμερίβερτ, θα ήθελα να σας παραπέμψω και στο ψήφισμα που εγκρίναμε πριν από μερικά χρόνια, με μεγάλη πλειοψηφία μάλιστα, ε, το ψήφισμα για το, για το λεγόμενο διαδικό σύστημα, dual system, ισορροπίας μεταξύ των ε, δημοσίων και ιδιωτικών ε, ΜΜΕ. Νομίζω ότι αυτό είναι θεμελιώδη σημασία ε, για να έχουμε έναν τέτοιο εξισορροπημένο πλουραλισμό στα ΜΜΕ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και, και χώρος για τις δημόσιες ε, επιχειρήσεις ε, για να κάνουν τη δουλειά τους ανεξάρτητα και αυτές. Και κατέστησα σαφές από την έρευνα που κάναμε τότε Εγώ ήρθα σε επαφή με πολλού τέτοιου οργανισμού και στην Ανατολική Ευρώπη και αλλού ότι υπάρχει πίεση από τι κυβερνήσει σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, ε, κάτι το οποίο καθιστά δύσκολη την ανεξάρτητη εργασία του. Ε, ε, πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σωστή ισορροπία Για λόγους λοιπόν ε, πλουραλισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και τα δημόσια ΜΜΕ. Και για όλες τις χώρες που θέλουν να προσχωρήσουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό ισχύει, αλλά και, για, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την προσχώρησή τους ε, συμφώνησαν ε, με την αρχή του σεβασμού ε, της, ελεύθερης, της ελευθεροτυπίας, της ελεύθερης έκφρασης και με όλα αυτά. Συμφώνησαν λοιπόν κατά την προσχώρησή τους. Δεν μπορούμε λοιπόν να το αμελήσουμε αυτό. Θα πρέπει να επιμείνουμε και να, να επενθυμίσουμε αυτά τα ζητήματα στις εθνικές αρχές αυτών των χωρών. Για το σημείο 2 Σίγουρα πρέπει να προσέξουμε οι δημόσιες αυτές επιχειρήσεις να μην βρίσκονται σε ένα είδους γκέτο και αυτό βέβαια έχει σχέση και με το ε, πρωτόκολλο του Άμστερνταμ, αλλά εδώ μιλάμε κυρίως για επικουρικότητα. Ταυτόχρονα η Επιτροπή πρόσφατα ε, εξέδωσε και κατευθυντήριες γραμμές για να μας δείξει τι ακριβώς μπορεί να κάνει ένα τέτοιο φορέα δημοσίου συμφέροντος ε, στο διαδίκτυο ή εκτός διαδικτύου. Και όλα αυτά βέβαια να τα έχουμε υπόψη. Για τα ιδιωτικά κανάλια, ιδιωτικοί φορεί, ε, βεβαίω είναι εξίσου σημαντική για την ε, διασφάλιση του πλουραλισμού στα ΜΜΕ. Οι ιδιωτικοί φορείς είναι ιδιωτικού δικαίου κατά κύριο λόγο και ιδιωτικών συμφερόντων. Εγώ για πολλά χρόνια εργάστηκα στον τομέα ε, των ε, ειδήσεων ε, και γι' αυτό λοιπόν ο συντάκτης και γι' αυτό θα πρέπει και οι συντάκτες να είναι σε θέση να, να προστατεύονται από την ηγεσία του μέσου, είτε αυτό είναι δημόσιο είτε ιδιωτικό και κατανοώ ότι η προστασία των συντακτών δεν είναι ποτέ απόλυτη, αλλά εφόσον θέτουμε ελάχιστα πρότυπα στην ε, Ευρώπη, θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Μετά για τα ιδιωτικά μέσα, μιλάμε και για τη συγκέντρωση των ΜΜΕ, το οποίο είναι το πιο σημαντικό σημείο σε αυτή την έκθεση. Ε, οι ισχυρέ επιχειρήσει σε ΜΜΕ. Εμεί δεν έχουμε πρόβλημα βεβαίω με αυτό, δεν είμαστε αντίθετοι. Είναι κάτι απαραίτητο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να δρούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δείτε τι συμβαίνει στι ε, ΗΠΑ και τη σχέση με την έκθεση του κυρίου Καβαντά. Είναι όμω πολύ σημαντικό και στην εθνική αγορά να υπάρχει επαρκή σε πλουραλισμό στα ΜΜΕ, να υπάρχουν αρκετά κανάλια, αν θέλετε, και φορεί σε ΜΜΕ Αυτά είναι ένα από τα κύρια καθήκοντα ε, της ομάδας υψηλού επίπεδου για, τα, για τον πλουραλισμό των ε, που έχει ε, διαμορφώσει η Επιτροπή. Θα θέλαμε να ακούσουμε και δύο λόγια από την Επιτροπή, να μας πείτε ακριβώς συμβαίνει, ε, τι συμβαίνει με την ενδιάμεση έκθεση, πότε να περιμένουμε την τελική έκθεση και ποια θα είναι τα κύρια σημεία, τα κύρια πορίσματα αυτής της έκθεσης. Έχουμε και το monitoring tool, το εργαλείο παρακολούθησης ε, του πλουραλισμού των ΜΜΕ, κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και μερικά χρόνια, που μας παρέχει ένα μαθηματικό μοντέλο, βάσει του οποίου μπορούμε να ε, μετρήσουμε το επίπεδο πλουραλισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, ανάλογα με διάφορους ε, παράγοντες. Και κατά τη χρήση του, χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, μπορούμε να έχουμε και μια πραγματική ε, ποσοτικοποιημένη εικόνα για το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα. Είναι κάτι που έχουμε στη διευθυνσία μας και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ακόμα περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Καβαντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι γρήγορος δεδομένης της ώρας και των περιορισμών της διερμηνίας. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον και ηρωνικό ταυτόχρονα. Το να μιλάμε σήμερα για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στην ιστορία μας ε, ε, για, είτε για την Ιταλία πριν από λίγα χρόνια, είτε για την Ουγγαρία τώρα και κάποιες άλλες χώρες ε, στη Γαλλία, υπάρχουν θεμελιώδη ζητήματα που τίθενται. Καταρχήν, οι θεσμοί ε, δυσκολεύονται να εφαρμόσουν όλες αυτές τις ε, γραπτές νομοθετικές αρχές. Θυμάστε τι συνέβη με, το χάρτ, με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το άτομο. Ε, χρειάζεται μια ισορροπία. Το με την άποψη του συναδέλφου που μίλησε πριν από λίγο. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, γιατί τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναπτυχθεί ε, αξιοθαύμαστα και το ρυθμιστικό πλαίσιο υπάρχει και λειτουργεί. Αλλά τα δημόσια μέσα ενημέρωσης πρέπει να πάρουν μια νέα ζωή, να αναζωογονηθούν. Γιατί εκείνα έχουν το κύριο δημοκρατικό καθήκον και όχι οι έμποροι του θεάματος οι έμποροι του θεάματος δεν ενδιαφέρονται ε, για, τους πολι... για τον πολίτη, για, τα... Για, το δικαίωμά τους, ε, για... Ε, για τα δικαιώματά τους. Καταρχήν, πρέπει να εφαρμόσουμε τα κείμενα, τα νομοθετικά που έχουμε στη διάθεσή μας, χωρίς επίοικια. Δεύτερον, να επαναφέρουμε μια οικονομική κυρίως ισορροπίας στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δεν είμαι ο μόνος ε, ο οποίος άκουσε το αίτημα για τη δημιουργία ενός νέου κρατικού τηλεοπτικού καναλιού, γιατί προφανώς υπάρχει μια τέτοια ανάγκη. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει και αυτός, αυτή η δίκαια κατανομή μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού. Τα ευρωπαϊκά κράτη δεν εφαρμόζουν πια δίκαια κατανομή γιατί δεν έχουν πόρους. Τώρα, όσον αφορά τα νομικά ζητήματα, ε, μένω κατάπληκτος που δεν έχουμε ακόμη σε όλες τις ε, ευρωπαϊκές χώρες ε, την υλοποίηση της Χάρτας των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Είναι, πρέπει οπωσδήποτε παντού να εφαρμόζεται ένα σύστημα προστασίας των δημοσιογράφων. Πολύ απέχουμε ακόμη από το να έχουμε εφαρμόσει τα πάντα με επιτυχία. Πολλά μένουν να γίνουν. Ε, επαναλαμβάνω, η επικουρικότητα, η αρχή της επικουρικότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι δυνατόν να συγχέουν την προπαγάνδα με την γενική υποχρέωση ε, που έχουν όλοι και κυρίως τα κράτη να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Λόκεγκάρντ, αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα το πρωί. Χαίρομαι για το γεγονό ότι υπάρχουν τόσα πολλά μέλη τη Επιτροπή μα που ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά και εγώ είμαι μεταξύ αυτών που θέλω να δείξω πραγματικά ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Συμφωνώ με την έννοια της δημόσιας υπηρεσίας που αναφέρθηκε προηγουμένως. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση σε κάτι το οποίο βρίσκεται στην έκθεση αυτή. Τα συμπεράσματα που έχουμε, στα οποία έχουμε καταλήξει σε πολλές εκθέσεις που έχουμε κάνει σε αυτή την Επιτροπή είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες, γιατί αυτές έχουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ποιότητα στις υπηρεσίες αυτές. Χρειάζεται λοιπόν μια ελευθερία πέραν των συνόρων σε ό,τι αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του δημοσιογράφου. Ένα άλλο θέμα είναι θέμα, το θέμα της χρηματοδότησης των δημοσίων υπηρεσιών. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα αυτά, στην ε, παρουσίαση στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση κτλ. Θα χαρώ λοιπόν πάρα πολύ να συζητήσω μαζί σας ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να με ποιους τρόπους μπορούμε να δώσουμε την, ε, τις πληροφορίες που χρειάζεται η Κομισιόν. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία να καταλήξουμε σε μορφές χρηματοδότησης που προωθούν την ε, ποιότητα της δημοσιογραφίας και δίνουν πραγματικά μια υπηρεσία στο ευρύ κοινό. Χρειάζεται φυσικά να υπάρχει και μια προστασία των πηγών των δημοσιογράφων, να υπάρξει η απαραίτητη απόσταση. Να εξασφαλίσουμε λοιπόν ένα μοντέλο Χρηματοδότηση το οποίο περιλαμβάνει την πλήρη ελευθερία για τους δημοσιογράφους να μπορέσουν να αποφασίσουν πώς θα εφαρμόσουν αυτό το μοντέλο. Είναι απαραίτητο να είναι γεγονός ότι εμείς θα έχουμε πράγματι εξασφαλίσει αυτή την ελευθερία των δημοσιογράφων. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Ο τελευταίος αυτό το γύρο συζήτησης, ο κύριος Τόκης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση. Με τα χαράς άκουσα τους συναδέλφους. Είναι κοινό τόπος ότι ε, όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει πλέον στην Ουγγαρία. Πρέπει λοιπόν ε, να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε την ελευθεροτυπία στην Ευρώπη. Αλλά να πω επίσης ότι υπάρχουν και πολλές παρανοήσεις ε, μαζί με άγνοια που οδήγησαν στις, ε, στην καταδίκη της κατάστασης στην Ουγγαρία. Κανείς δεν γνωρίζει ότι στην Ουγγαρία μετά την ε, περίοδο την περίοδο μετά τον, τον κομμουνισμό υπήρξε μια τεράστια αλλαγή στην εξουσία και έτσι λειτουργεί πλέον ο τύπος, ο φιλελεύθερος τύπος και αυτό έχει αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική μετάβαση που ξεκίνησε το 1989. Δεν ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η μετάβαση. Στη Δύση τα βλέπουμε λίγο ασπρόμαυρα τα πράγματα ως προς αυτό το θέμα. Η κατάσταση όμως είναι διαφορετική στην πραγματικότητα. δεν ε, μπορούμε να φτάσουμε τον ε, ακραίο φιλελευθερισμό βάση της ελευθεροτυπίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε και την κατάσταση στη συγκεκριμένη χώρα ε, μετά το, την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος κτλ. Πέρα από, τα, από την Ουγγαρία, για παράδειγμα στη Ρουμανία, βλέπουμε πολύ μεγάλες οικονομικές δυνάμεις ε, με τεράστια πολιτικά συμφέροντα. Και εκείνοι έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, στο χέρι. Ε, χειραγωγούν λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους Ρουμάνους πολίτες ως συνέπεια. εδώ πρέπει να μιλούμε για την πραγματική ανεξαρτησία των ΜΜΕ. Σε πολλέ περιπτώσεις υπάρχει και εξαγορά των ΜΜΕ και ω εκ τούτου πολλές ευθύνε. Πολυεπίπεδη λοιπόν η κατάσταση εδώ. Γιατί δεν θέλουμε να τρομοκρατούμε ή μάλλον να, διαμορφώσουν, να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα τρομοκρατία μέσω ε, των μέσων μαζική ενημέρωση. Ευχαριστώ κύριε Τόκε. Και τώρα α δούμε αν υπάρχει εκπροσώπηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ο κύριο Τρέτενμπέιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε αναφερθεί ήδη μια σειρά από δραστηριότητες που συνοδεύουν τις τόσο σημαντικές αυτές τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στο Κοινοβούλιο και που βρίσκονται και επίσης στην, στον τη της μέρης της Κομισιόν να υποστηρίξουν τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης για μια δημοκρατική κοινωνία. Ο κύριος Μπέλετ έθεσε το ερώτημα πού βρίσκεται η επεξεργασία από την ομάδα εργασίας ε, αυτή η ομάδα εργασία με επικεφαλή τον κύριο Φράιμπεργα, την κυρία Φράιμπεργα, την πρώην πρόεδρο της, ε, έχει ήδη συνεδριάσει κάποιες φορές και θα συζητήσει και στο μέλλον. Εξετάζει τις απειλές προς τα μέσα ενημέρωση σε ό,τι αφορά τον πλουραλισμό και την ελευθερία και θα κάνει συστάσεις στην τελική της έκθεση σε όλους τους εμπλεκόμενους και στο Συμβούλιο και στα κρατημέλη και στην Κομισιόν αντιμετωπίζοντας και τα παραδοσιακά και τα νέα μέσα και καλύπτοντας ένα σύνολο προβλημάτων από περιορισμούς μέχρι ελευθερία έκφρασης και για να παρουσιάσει προτάσεις για το πώς μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη λογοδοσία, εμπιστοσύνη, ε, προστασία των πηγών των δημοσιογράφων κτλ η ομάδα αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να καλύψει όλο αυτό το ευρύ πεδίο και ζήτησε να υπάρξει μια παράταση της εργασίας της ομάδας. Προβλεπόταν μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 η ομάδα αυτή να δώσει την έκθεσή της. Τώρα όμως η γενική εντύπωση είναι ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο και το νωρίτερο θα είναι στο τέλος του 2012 που θα μπορούσε να προκύψει μια έκθεση της ομάδας και δεν προβλέπεται βέβαια ενδιάμεση έκθεση. Υπάρχουν και άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες εν εξελίξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Και εμείς υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενός κέντρου για την πολυμορφία και την ελευθερία των μέσων στο, στην έδρα Ρόμπερ Σούμαν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Ο στόχος είναι να υπάρξει και μια σειρά από έγγραφα πολιτικής που θα προετοιμάσουν ε, την συνολική λήψη απόφασης και θα προσδιορίσουν τι μπορεί να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά. Και στο περιθώριο αυτών υπάρχει η ομάδα Φοντήλο η οποία εξετάζει το σύνολο αυτών των θεμάτων νέα μέσα εξελίξεις στα μέσα ενημέρωσης, διαταραχές στην ελευθερία των έντυπων μέσων κτλ. Πώς μπορούμε να τα υποστηρίξουμε όλα αυτά από την ευρωπαϊκή πλευρά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σε σχέση με τις ε, συστάσεις που αναφέρατε. Έχω ένα ερώτημα όμως. Όταν προτείνεται εδώ να δοθεί έμφαση στο παιδαγωγικό μοντέλο των κρατικών μέσων οι εμπορικές δραστηριότητες των δημοσίων μέσων θα είναι μονάχα συμπληρωματικέ προς την ε, πρόθεση των πολιτιστικών και άλλων αρχών. Και η κυρία Κάμεφερτ ρώτησε πώς συνδέεται αυτό με το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφήνει στα κράτη-μέλη να καθορίσουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μέσων ενημέρωσης. Γιατί οι εμπορικές τους δραστηριότητες γιατί θα πρέπει να περιορίζονται στην αποστολή δημόσιας υπηρεσίας των ε, ε, των μέσων αυτών. Αυτό φαίνεται ότι δημιουργεί κάποια σύγχυση. Ευχαριστώ την Επιτροπή και για τα τελικά συμπεράσματα ο εισηγητής Νεγκάσκη. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Σημείωσα τρία πράγματα τα οποία οποία επισημάνατε επενειλημμένως και τα οποία θα επανεξετάσει στο τελικό στάδιο της έκθεσης. Είχα μόνο 1.800 χαρακτήρες στην έκθεσή μου. Ε, εσείς αναφερθήκατε κυρίως στην ελευθερία, στον πλουραλισμό, σε αυτά τα σημεία και είπατε ότι αυτή πρέπει να είναι η βάση του των μελλοντικών μας εργασιών. Πολύ σύντομα να, παρα... να στην Επιτροπή. Πρόθεσή μου ήταν να αναγνωρίσουμε ότι τα δημόσια, τα, κρατικά μέσα που μπορούν να έχουν και εμπορική δραστηριότητα μέσω διαφημίσεων ή άλλων στοιχείων που δεν αποτελούν ε, αναπόσπαστο τμήμα της αποστολής τους πρέπει να, να λειτουργούν συμπληρωματικά. Η αποστολή τους είναι η ορθή και αντικειμενική ενημέρωση του κοινού. Ο στόχος λοιπόν ήταν να δούμε τι ακριβώς κάνουν τα, δημόσια μέσα για να συγκεντρώσουν πόρους και ότι αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να είναι συμπληρωματικές και να μην παρεμποδίζουν την ε, αρχική αποστολή αυτών των μέσων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μιγκάσκε. Στο σημείο αυτό σας θυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 12η Απριλίου, 12 η ώρα και θα ψηφίσουμε το Μάιο. Εδώ θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα στις 3 έχουμε μια δημόσια ακρόαση για την διαμόρφωση του μελλοντικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και τη νεολαία. Και θα ακολουθήσει η συνδιάσκεψη ε, των εισηγητών. Των συντονιστών, με συγχωρείτε.